Σα Σας καλωσορίζω θερμά στη σημερινή συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Ε, καλωσορίζω τους ε, συναδέρφους, ε, τους εκπροσώπους ε, της ε, Κομισιόν και του Συμβουλίου, τους ακροατές μας που είναι παρόντες σήμερα. Σας καλωσορίζω λοιπόν θερμά στην συνεδρίαση της Επιτροπής μας. ιδιαίτερα θέλω να καλωσορίσω ένα μέλος του Σουηδικού Κοινοβουλίου που εργάζεται σε θέματα ισότητας ε, που βρίσκεται εδώ σήμερα για να δει πώς χειριζόμαστε τα θέματα ισότητα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, καλώς ήρθατε λοιπόν. Έχουμε και άλλους ε, επισκέπτε από τη Σουηδία. Από το Ρινταχόλμ και τη Βίσλαντα, σας καλωσορίζω και εσάς. Ε, ήρθατε εδώ για να ακούσετε την συνεδρίαση της Επιτροπής μας σήμερα. Ε, πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Ε, έχω πρόταση για προσθήκη στην ημερήσια διάταξη. Συζήτηση και υιοθέτηση, έγκριση μιας προφορικής ερώτησης προς την Κομισιόν όσον αφορά την ε, παρακολούθηση της συνέχειας που έχει να κάνει με ένα καταστατικό για τα δικαιώματα των γυναικών. 13α ε, ε, θα είναι το θέμα αυτό στη μερίσια διάταξη. Έχει ζητήσει το λόγο η κυρία Πάρα. Ε, Ευχαριστώ. Αύριο θα έχουμε ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο, την Vivian Redding. Και επειδή έχουμε αμέσως μετά συνάντηση των συντονιστών, προτείνω να αποφασίσουμε στη συνεδρίαση αυτή των συντονιστών η χάρτα των δικαιωμάτων των γυναικών τι μέλλον θέλουμε να έχει. Δεδομένου ότι τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι διαφορετικά και δεν θα θέλω να λάβουμε απόφαση σήμερα για κάτι ε, για το οποίο θα μπορέσουμε να διαμορφώσουμε άποψη αύριο μόνο. Οπότε α μην προσθέσουμε αυτό το θέμα στη σημερινή ημερήσια διάταξη, αλλά να το αποφασίσουμε αύριο στι συνεδρίε των συντονιστών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπάουερ. Κυρία Κορνέλισεν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι έχει δίκιο η κυρία Μπάουερ. Όταν λέει ότι πρέπει να το συζητήσουμε αύριο στους συντονιστές. Το τι θα κάνουμε δηλαδή αφού θα το συζητήσουμε και με την ε, κυρία Ρέντινγκ. Εγώ ως συντονίστρια θα ήθελα να ακούσω μερικές από τις απόψεις ε, άλλων ε, στην Επιτροπή μας για να μπορούσα να το λάβω αυτό υπόψη στις συζητήσεις των συντονιστών αύριο. Ευχαριστώ κυρία Τόμσεν. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συζητήσουμε τον χάρτη δικαιωμάτων των γυναικών ε, στην Επιτροπή μας με την κυρία Ρέντινγκ ως εκπρόσωπο της Κομισιόν. Διότι όταν ο κύριος ε, Μπαρόσο βρισκόταν στην αντιπροσωπεία ΠΕΣ ε, στην εκστρατεία για την επανεκλογή του στην Επιτροπή, τον ρωτήσαμε αν τον εκλέξουμε, εάν θα παρουσιάσει χάρτη δικαιωμάτων των γυναικών και το υποσχέθηκε. Είπε ότι στο όνομα της Επιτροπής θα παρουσιάσει χάρτη δικαιωμάτων των γυναικών. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τον χάρτη αυτόν, διότι ε, το προσυπογράφει μόνο η Κομισιόν και όχι όλα τα θεσμικά όργανα της Επιτροπής. Δεν έχει τη μορφή που θέλουμε, γι' αυτό επιμένω να γίνει η συζήτηση για το χάρτη δικαιωμάτων των γυναικών. Ευχαριστώ. Η κυρία Παρβάνοβα, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που είπαν ήδη οι συνάδελφοι, αλλά νομίζω ότι η δέσμευση των τριών επιτρόπων και του Προέδρου κατά τη διάρκεια του πρωινού μας ήταν ε, κάτι πολύ διαφορετικό από το αποτέλεσμα που βλέπουμε και είναι πολύ σημαντικό να έχουμε τη συζήτηση αυτή. Όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας της Κομισιόν, δεν βλέπουμε πουθενά ε, κάτι για την ε, βία όσον αφορά τα φύλλα και πιστεύω ότι θα πρέπει να του πιέσουμε για να έχουμε σαφή απάντηση στο θέμα αυτό. Δεν είμαι ικανοποιημένη με την πρόταση και πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρξει συζήτηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Παρβάνοβα, κυρία Γιανακουδάκη. Yes. Um, yes, it's a very important issue, this charter. Ναι, είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό του χάρτη και ανησυχώ λίγο ότι θα συζητήσουμε κάτι Πρωτού ακούσουμε τι ε, έχει να πει η Ρέντινγκ και αν έχουν κάνει κάτι. Μήπως θα ήταν καλύτερα λοιπόν να περιμένουμε ε, να δούμε πρώτα τι θα γίνει, ε, να δούμε προς, τα πού πηγαίνουν στην αυριανή συνεδρίαση και μετά να συζητήσουμε. Προτείνω δηλαδή να περιμένουμε να δούμε πρώτα τι έχει να μας πει η κυρία Ρέντινγκ. Ευχαριστώ κυρία Φιγερέδο. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τις συναδέλφους υπό την έννοια ότι θα πρέπει να γίνει μια διασάφηση αυτού του ζητήματος διότι μας υποσχέθηκαν μια συζήτηση η οποία δεν ε, επιβεβαιώθηκε και γι' αυτό ακριβώς θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Ξέρω ότι σήμερα το πρωί θα παρευρεθεί εδώ η κυρία Ρέντινγκ και θα μιλήσουμε μαζί της επί του θέματος, αλλά θα πρέπει να λάβουμε θέση. Και γι' αυτό νομίζω ότι η διάσκεψη, αλλά και η Επιτροπή, καθώς και η δήλωση της ε, Προέδρου, θα πρέπει να οδηγήσει στην επαύξηση της σημερινής διάταξης με άλλο ένα σημείο. Νομίζω λοιπόν ότι ή πριν ή μετά την ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Ρέντιν θα πρέπει να ανταλλάξουμε απόψεις για τις δράσεις που θα πρέπει να αναπτύξουμε ε, γύρω από αυτό το ζήτημα μαζί με την Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Φιγκερέιδο, κυρία Σαμπόρσκα. E, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να τονίσω ότι η κυρία Μπάουερ δεν θέλει να αμφισβητήσει το αν θα πρέπει η Επιτροπή μας να συζητήσει η Επιτροπή μας το θέμα του χάρτη των ε, δικαιωμάτων των γυναικών. Ε, η κυρία Μπάουερ μίλησε μόνο για το χρονοδιάγραμμα. Πότε θα πρέπει να θέσουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη. Εγώ πιστεύω ότι η ημερήσια διάταξη όπως προτείνεται, δηλαδή αύριο να έχουμε τη συζήτηση με την κυρία Ρέντινγκ και να γίνει και μετά η συνεδρία των συντονιστών και λογική συνέπεια να είναι οι συντονιστές των πολιτικών ομάδων να συζητήσουν το χάρτη των δικαιωμάτων των γυναικών. Βρισκόμαστε στην αρχή της ε, νομοθετικής θητείας και δεν χάνουμε χρόνο εάν θέσουμε το θέμα αυτό στη μέση διάταξη του επόμενου μήνα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Σαπόσκα. Η κυρία Μπάουερ. Ε, I have nothing, nothing to add. Δεν έχω τίποτε να προσθέσω. απλώ να τονίσω ότι δεν έχω πρόβλημα να κάνουμε τη συζήτηση για το θέμα αυτό. Το πρόβλημα είναι το χρονοδιάγραμμα. Δεν υπάρχει λόγος να βιαζόμαστε. Να ακούσουμε πρώτα τη συμβολή της κυρίας Ρέντινγκ για το θέμα και μετά. Ευχαριστώ κυρία Μωρέν. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με την δεύτερη παρέμβαση της κυρίας Μπάουερ. Ακούγοντας τις συναδέλφους θα έλεγα ότι όλοι συμφωνούν με την ιδέα ότι το θέμα αυτό είναι σημαντικό και ότι θέλουμε να επενδύσουμε σε αυτό, να προβληματιστούμε αλλά άλλο η ταχύτητα και άλλο η βιασύνη. Και το, πω, το, το ότι θα έρθει εδώ η κυρία Ρέντινγκ είναι πολύ σημαντικό. Είναι σημαντικό να την ακούσουμε πριν να είμαστε σε θέση να προτείνουμε κάτι, να τοποθετηθούμε. Βάσει μιας ε, συζήτησης για την οποία θα έχουμε ήδη λάβει κάποια στοιχεία. Συμφωνώ λοιπόν με την ε, σοφία άποψη της ε, τελευταίας παρέμβασης κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τις απόψεις που εκφράσατε. Θα ήθελα απλά να σας θυμίσω ότι συζητάμε την προσθήκη ενός θέματος στην ημερήσια διάταξη κατά την αυριανή συνεδρίαση. Πρόκειται για προφορική ερώτηση μετά τη συνάντηση που θα έχουμε στις 9 με 10 η ώρα αύριο το πρωί με την Επίτροπο Ρέντινγκ. Υπάρχουν από ό,τι κατάλαβα διαφορετικέ απόψει σχετικά με το αν θα πρέπει να θέσουμε το θέμα αυτό στην ημερήσια διάταξη αύριο ή όχι. Θα ήθελα επίση να, να σα θυμίσω ότι πρόκειται απλά για προφορική ερώτηση. Αργότερα θα συζητήσουμε ενδεχόμενο κείμενο ψηφίσματος. Πρόκειται απλά λοιπόν για προφορική ερώτηση που έχει σκοπό να τεθεί το ερώτημα προς την Κομισιόν τι παρακολούθηση της συνέχεια θα γίνει όσον αφορά το χάρτη δικαιωμάτων των γυναικών. Καθότι όμως υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, διστάμενες απόψεις, προτείνω να ψηφίσουμε. Εάν θα πρέπει να θέσουμε το θέμα στην ημερήσια διάταξη της αυριανής συνεδρίασης ή όχι. Όσοι πιστεύουν ότι θα πρέπει να προσθέσουμε ένα σημείο 13α στην αυριανή ημερήσια διάταξη, παρακαλώ σηκώστε το χέρι σας. Δηλαδή, συμφωνείτε να συζητηθεί το θέμα. Ποιος είναι κατά. Αποχές. Καμία αποχή. Τέσσερις, ε, συγγνώμη, δέκα είναι υπέρ του να τεθεί το θέμα στη μερίσια διάταξη αύριο και οχτώ ψήφισαν κατά. Το αποτέλεσμα είναι ότι θα θέσουμε το θέμα στην ημερήσια διάταξη αύριο. Ε, θα είναι το σημείο 13α. Άλλες τροποποιήσεις στην ημερήσια διάταξη. Η κυρία Τόμσεν ζήτησε το θέμα της που είναι η ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργία θέσεων εργασία στο πλαίσιο μια νέα βιώσιμη οικονομία. να, να ε, τεθεί στο σημείο 4 τη ε, ημερησία διάταξη, να αλλάξουμε δηλαδή θέση με την έκθεση για την κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών που ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων. Μπορούμε να το κάνουν αυτό. Έτσι λοιπόν έχουμε εγκρίνει την ε, ημερήσια διάταξη για τη σημερινή συνεδρίαση. Σημείο 3. Έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων στις 23 Φεβρουαρίου, 7 Απριλίου και τα πρακτικά βρίσκονται στα έγγραφά σας. Εάν δεν καταγραφούν αντιρρήσεις μέχρι το πέρας της συνεδρίασης, θα θεωρηθεί ότι έχουν εγκριθεί τα πρακτικά και έτσι προχωράμε αμέσως ε, στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης με την τροποποίηση που κάναμε. Το θέμα αυτό αφορά την ανάπτυξη του δυναμικού δημιουργίας θέσεων εργασίας στο πλαίσιο μιας νέας βιώσιμης οικονομίας. Στις 30 ε, Νοεμβρίου πέρσι οι συντονιστές συμφώνησαν να εκπονηθεί συνεδρία, ε, έκθεση προς την γνωμοδότηση προς την Επιτροπή αν, ε, Απασχόλησης. Η κυρία Τόμσεν ορίστηκε η συγγήτρια και της δίνω το λόγο για να ε, παρουσιάσει τη σημερινή συζήτηση. Παρακαλώ κυρία Τόμσεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Βρισκόμαστε σε κατάσταση κρίσης στην Ευρώπη. Και θέλουμε η οικονομία μας και η αγορά εργασίας ε, που θα υπάρχει όταν ολοκληρωθεί η... όταν τελειώσει η κρίση είναι διαφορετική από αυτήν που είχαμε. Και διακόπτει ομιλήτρια. No Danish translation today, so I'll try in English. Δεν έχει δανέζικη διερμηνία σήμερα, θα τα πω αγγλικά λοιπόν. New economy when we will get through the... Μετά την ε, κρίση θα, δούμε, θα περάσουμε σε μια νέα οικονομία και η ευρωπαϊκή οικονομία δεν θα είναι η ίδια που ήταν πριν την κρίση και αντί να επικεντρωθούμε στις περικοπές ε, στα μέτρα ισότητας ε, και στην απασχόληση που συνήθως πλήττουν τις γυναίκες καθότι το 75% ε, των απασχολούμενων στον δημόσιο τομέα είναι γυναίκες. Πιστεύω λοιπόν ότι θα πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία και είναι ζωτική σημασία αυτό. Είναι λοιπόν ζωτική σημασία να χρησιμοποιήσουμε την οικονομική κρίση για να ε, εξαλείψουμε τα εμπόδια στην ισότητα στην ε, αγορά εργασίας, διότι η νέα οικονομία θα βασίζεται σε μια πράσινη οικονομία και σε μια οικονομία που θα βασίζεται στην τεχνολογία της πληροφορικής. Τώρα όταν αναλύουμε την κατάσταση στην, ε, στον τομέα της ενέργειας και του περιβάλλοντος βλέπουμε το 80 με 85% ε, των θέσεων απασχόλησης το κατέχουν άντρες. Και αν ε, εξετάσουμε τα στοιχεία από την αγορά εργασίας, είναι πολύ σημαντικό οι γυναίκες να μπουν στην αγορά εργασίας σε όλα τα επίπεδα στη νέα οικονομία, στο νέο πράσινο τομέα. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να παρέχεται εκπαίδευση, τεχνική κατάρτιση στις γυναίκες και θα πρέπει εδώ να συμμετάσχει και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Από ό,τι με ενημερώνουν μόνο το 10% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου χρησιμοποιήθηκαν κατά την προηγούμενη περίοδο στην κατάρτιση γυναικών. Και πιστεύω ότι πραγματικά θα πρέπει να καταβάλουμε προσπάθεια στον τομέα αυτών. Επίσης θα πρέπει να φροντίσουμε οι γυναίκες να μπορούν να έχουν σταδιοδρομίες ε, στους νέους τομείς ε, χαμηλών εκπομπών ε, διοξιδίου του άνθρακα στην οικονομία. Σημαντικό είναι να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των γυναικών στις θέσεις απασχόλησης αυτές, καθώς και τα δικαιώματα των εργαζομένων στους νέους αυτούς τομείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Τόμσεν. Ε, δίνω το λόγο στους συναδέλφους για να ακούσουμε τις απόψεις τους. Η κυρία Κορνέλησεν, παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ διάβασα με πολύ χαρά την έκθεση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επίκαιρη, πάρα πολύ σημαντική γιατί δουλεύουμε πολύ σκληρά για την ε, Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 ε, και ε, βλέπουμε και τους στόχους που έχουμε για την απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα επόμενα 10 χρόνια και επομένως είναι εξαιρετική σημασία η πτυχή της ισότητας των φύλων να συμπεριληφθεί στην όλη διαδικασία. Αρχίζουμε σιγά σιγά να ασχολούμαστε με τις κατευθυντήριες γραμμές απασχόλησης και πρέπει η πτυχή να ληφθεί υπόψη και σε αυτόν τον τομέα. Και θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την έκθεση αυτή ως συμβολή σε αυτό. Η κυρία Σρέτερη, η πράσινη συνάδελφος, ε, είναι η συγγήτρια της ε, Επιτροπής Απασχόλησης για αυτό το θέμα και ήταν και μέλος Επιτροπής Γυναικών και χαίρομαι όλος ιδιαίτερος που ισχύει αυτό, γιατί αυτό σημαίνει ότι gender mainstreaming γίνεται και μεταξύ ημών. Όσον αφορά τώρα τη διαβίου μάθηση και την εκπαίδευση ώστε να εξασφαλίσουμε ότι δεν μένουν οι γυναίκες πίσω σε μια οικονομία ε, με χαμηλές εκπομπές άνθρακα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό θα μπορέσουμε έτσι να μειώσουμε και τις ανισότητες στις αμοιβέ μεταξύ ανδρών και γυναικών. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020 για τις κατευθυντήριες γραμμές για την ε, απασχόληση είναι ότι δεν έχει πρικοδοτηθεί με τίποτε ε, η συγκεκριμένη διαδικασία. Και αυτό είναι σημαντικό να το αναφέρουμε. Το, η επιχειρηματικότητα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Βέβαια το διάβασα υπό το φως των ε, τροπολογιών που ενδεχομένως να, το, να βελτιώσουν τα συγκεκριμένα σημεία. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Νομίζω ότι μπορούμε να βελτιωθούμε όσον αφορά στου τομεί όπου κυριαρχούν οι άντρε για να συγκεράσουμε οικογενειακό και επαγγελματικό βίο και να αλλάξουμε την κουλτούρα των γραφείων. Επίση, ε, μια, χαμη... μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα δεν είναι μόνο υψηλή τεχνολογίας, προηγμένη τεχνολογίας ε, για τους μηχανικούς, ε, αλλά έχει να κάνει γενικότερα με τη θεώρηση της υφόρου οικονομία που αφορά όλους τους τομείς. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω τη γύρανση της κοινωνίας, γιατί βρισκόμαστε σε μία δεκαετία όπου μπορεί να έχουμε αηφόρο οικονομία, αλλά θα έχουμε και γυράσκοντα ενεργό πληθυσμό. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι κάθε γυναίκα που μπορεί να εργαστεί, τη χρειαζόμαστε στο εργατικό δυναμικό μας και πρέπει να καταστήσουμε την αγορά εργασίας ελκυστική για τις γυναίκες αυτές. Είμαι σκιώδης εισηγήτρια για τις κατευθυντήριες γραμμές ε, το, της απασχόλησης ε, στην Επιτροπή ε, απασχόλησης ε, και θα ήθελα πραγματικά να ακούσω τι έχουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι να πούνε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Κονέλης. Είναι η κυρία Σαπόσκα, παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Τόμσεν για, την, για το σχέδιο γνωμοδότησης που συνέταξε. Πιστεύω ότι η Στρατηγική Ευρωπαϊκή Ένωση 2020 είναι το πλαίσιο πολιτικής για τα, την επόμενη δεκαετία και έχει άμεση σχέση με την έκθεση που συζητούμε αυτή τη στιγμή. Είναι η στιγμή να ε, υποβάλουμε τις ευχές μας και τις, επιθυμίες μας. Ε, κυρίως για την πολιτική των γυναικών ε, στην αγορά εργασίας. Υπάρχει μεγάλος ε, κίνδυνος ε, διατήρησης των προηγούμενων πολιτικών απασχόλησης και επειδή βρισκόμαστε σε κρίση, οι αρχές πρέπει να αναθεωρηθούν. Θα ήθελα να αναφερθώ στην τροπολογία της κυρίας Γκαρσία Πέρες, η οποία πολύ μου αρέσει η κυρία Πέρες ε, στην τροπολογία της αναφέρει ότι δεν μπορούμε πια να παραμείνουμε κολλημένοι σε αρχές ε, που δεν έχουν κανένα, καμία ουσία. Να θέλουμε αηφόρο οικονομία με ε, καταμερισμό εργασίας εντελώς παροχημένο σε σχέση με τη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας Χρειαζόμαστε νέα μοντέλα που βασίζονται στην καινοτομία και τη γνώση. Πιστεύω επίσης ότι και η υπερβολική νομοθεσία δεν βελτιώνει πάντοτε την καθημερινή ζωή. Η αποτυχία της στρατηγικής της Λισαβόνας, οι απαιτήσει ε, της ε, δημοκρατικής πρόκλησης ε, ουσιαστικά μας καλούν μαζί με την κατάσταση της γυναίκας ε, στην οικογενειακή τη ζωή, τη φτώχεια των γυναικών, μας καλεί λοιπόν να ε, ασχοληθούμε πιο προσεκτικά με τα προβλήματα της γυναίκας και στην καθημερινή της ζωή και δεν πρέπει να ξεχνούμε στην έκθεση την αναγνώριση της ε, άτυπης εργασίας και τον, την, τα εξαρτώμενα πρόσωπα. Ευχαριστώ κυρία Σαπόρσκα. Η κυρία Αντιπρόεδρος Μωρέν έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω όλους όσους ε, είπαν την άποψή τους στην κυρία Τόμσεν ε, για την ε, δουλειά της. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό, όπως και η κυρία Κορ... Ε, είμαι και εγώ στην Επιτροπή Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων και βλέπουμε ότι με την έκθεση αυτή ασχολούμαστε με ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, ένα πολύ σημαντικό ζήτημα επί του οποίου πρέπει να κάνουμε μία τομή, γιατί η κρίση ε, καθιστά πιο ευάλωτες ε, τις γυναίκες, τέλος πάντων την κατάσταση των ε, γυναικών που ήδη βρίσκονταν σε άνεση θέση με τους υπόλοιπου στην κοινωνία. Σήμερα οι νέες γυναίκες ε, έχουν πολλά διπλώματα, έχουν πολλά προσόντα, το να επιτύχουν καλύτερα στις σπουδές τους ε, ε, δεν σημαίνει υποχρεωτικά ότι αυτό μειώνει τις ε, μισθολογικές διαφορές και συχνά έχουν πρόσκαιρη απασχόληση και φτάνουν οι γυναίκες στο τέλος επαγγελματικής του ζωής πολύ πιο φτωχές από τους άνδρες. Πέντε χρόνια χρειάζονται για τη γυναίκα να φτάσει το μισθό που ένας άντρας παίρνει σε τέσσερα χρόνια. Οπότε πρέπει σε αυτήν την έκθεση και ε, στο πλαίσιο της εργασίας Επιτροπής Απασχόλησης Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει πραγματικά να δραστηριοποιηθούμε. Πρέπει να επικεντρώσουμε την προσπάθειά μας όσον αφορά τη μείωση των μισθολογικών διαφορών. Δεύτερον, ε, την συμφιλίωση, τους μηχανισμούς συμφιλίωσης μεταξύ οικογενειακού και επαγγελματικού βίου, γιατί πάντοτε οι γυναίκες ε, θα έχουν να αντιμετωπίσουν ε, τέτοιου είδους ε, εμπόδια και αν κάνουμε προσπάθειες για τις νέες γυναίκες και την εκπαίδευσή τους πρέπει να, τους, να τις βοηθήσουμε κιόλας να συμφιλιώσουν την επαγγελματική και την οικογενειακή τους ζωή. Πρέπει επίσης να βελτιώσουμε, να αυξήσουμε το μερίδιο του κοινωνικού ταμείου που είναι αφιερωμένο στη μείωση των διαφορών ε, μεταξύ του επαγγελματικού βίου των γυναικών και των ανδρών, ενισχύοντας τη διαβίου εκπαίδευση και κατάρτιση. Είναι καθήκον μας ε, να θέσουμε εδώ ένα νέο στόχο, και βέβαια υπάρχει και ένα τέταρτο και σημαντικό σημείο, το οποίο, το επίσης μου φαίνεται λοιπόν πολύ σημαντικό, είναι να λάβουμε υπόψη μας ε, και το γεγονός ότι ε, το προσδόκιμο ζωής είναι πλέον μεγαλύτερο. Υπάρχουν νέες, ε, υπάρχει νέα κοινωνική εργασία, νέες μορφές, την οποία επίσης πρέπει να τονίσουμε, προς όλων και πρέπει πραγματικά να ε, αφοσιωθούμε σε αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Μωρένη, κυρία Μπάουερ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα απλά, επειδή όλα όσα ήθελα να πω υπόθηκαν, ε, θα ήθελα να πω πώς εκτιμώ την προσέγγιση της κυρία Τόμσεν, διότι Είμαι βεβαία ότι η μελλοντική οικονομία δεν θα είναι η ίδια με αυτήν που είχαμε πριν την κρίση. Είναι απαραίτητο να έχουμε κατά νου ότι όλες οι προβλέψεις λένε ότι δεν θα αντικατασταθούν όλες οι χαμένες θέσεις απασχόλησης. οι νέες θέσεις απασχόληση που θα δημιουργηθούν θα δημιουργηθούν κυρίως σε δύο περιθωριακές θέσεις του προγράμματος απασχόλησης, δηλαδή άτομα ε, χαμηλής εξειδίκευσης στον τομέα των υπηρεσιών και άτομα υψηλής ε, εξειδίκευσης, κυρίως ε, για νέες τεχνολογίες και νέες δεξιότητες. είναι απαραίτητο να τονίσουμε και να έχουμε κατά νου ότι η ιδέα της Ατζέντας 2020 είναι να αυξήσουμε με ποσόστοση την απασχόληση των γυναικών από 60 σε 75%. Αυτό σημαίνει ότι αυτό είναι απολύτως αδύνατον, διότι θα χρειαστούν αρκετά διαφορετικά βήματα στον, ε, στη διαδικασία της συνδιαλλαγής. Δεν θα μπορέσουμε να αποφύγουμε το θέμα αυτό στη γνωμοδότηση αυτή. Αυτό ήθελα να προσθέσω όσον αφορά τη γνωμοδότηση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τελευταία ομιλήτρια είναι η κυρία Κώστα προτού να δώσουμε το λόγο στην κυρία Τόμσεν για την τελική παρέμβαση. Παρακαλώ, κυρία Κώστα. Ευχαριστώ. Εκτίμησα ιδιαίτερα την, πρόσταση, την πρόταση έκθεση της κυρίας Τόμσον και νομίζω ότι έχει σταθεί σε βασικούς πυρήνες. Θα ήθελα να θίξω δύο ζητήματα που ίσως μπορούν να εμβαθυνθούν. Μιλάμε ότι για το θέμα της οικονομικής βιωσιμότητας. Ε, μιλάμε για βιωσιμότητα και κοινωνική και περιβαλλοντική. Αυτά τα δύο σκέλη μπορούν να συνδεθούν, διότι έτσι μπορούμε να λάβουμε υπόψη και τον παλαιό τρόπο παραγωγικών μηχανισμών, αλλά και μία εργασία η οποία να οδηγεί περισσότερο στην ε, ευελιξασφάλεια και να είναι φιλική προς την οικογένεια. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη την κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης, η οποία θα πρέπει να ξανασκεφτεί τα σχήματα εργασίας. Δηλαδή μια δράση πιο φιλική προς τις γυναίκες και προς την οικογένεια. Συμφωνώ με το θέμα της χρήσης του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ήμουνα υπεύθυνη στην περιφέρειά μου για πέντε χρόνια σε αυτό το τομέα, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθεί καλύτερα το ΕΚΤ. Θα πρέπει λοιπόν να μας απασχολήσει και με την Επιτροπή Ρέτζο, γιατί από του χρόνου θα έχουμε νέες κατευθυντήριες γραμμές για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το mainstreaming, αλλά ίσως ήταν ένα άλλο στο κοινωνικό τομέα για να μην εστιάσουμε πια την προσοχή μας στις γυναίκες. Μιλάμε για ένα 10% στοχοθέτηση. Ίσως θα μπορούσαμε να συνδυάσουμε τις δύο προσεγγίσεις έτσι ώστε να τα δούμε όλα αυτά υπό μία νέα προοπτική με βάση τους απότερους στόχους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Ευχαριστώ κύριε Κώστα. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για το μέλλον. Το βλέπουμε ε, και στον αριθμό των βουλευτών που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Έχω άλλους δύο στην ημερησία διάταξη. Πρώτα η κυρία Σέσκοβα, παρακαλώ. Ε, αυτό που έχει σημασία είναι να λάβουμε υπόψη ότι ο κοινωνικός τομέας... Δυστυχώ ε, Δυστυχώς ε, δεν μπορεί να γίνει διερμηνία από τη γλώσσα αυτή. Συγγνώμη, δεν υπάρχει διερμηνία. Είναι δυνατόν να μιλήσετε αγγλικά, γαλλικά. Ωραία, θα μιλήσω αγγλικά, αγγλικά, αλλά είναι πολύ διαφορετικό να μπορεί κανείς να εκφραστεί στη μητρική του γλώσσα. Άκουσα ε, διερμηνή από τα σλοβακικά ή έτσι μου φάνηκε. Το ζήτησε η βοηθός μου, αλλά σας έχουμε ζητήσει εδώ και ένα χρόνο να έχω διερμηνία. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να πω τα εξής. Μας ενδιαφέρει η ισότητα. Αυτό είναι κάτι πολύ θετικό. Ζητώ συγγνώμη, αλλά νομίζω ότι ορισμένες φορές δεν λαμβάνουμε υπόψη τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες. γιατί θεωρούμε ότι δεν χρειάζονται αυτή την προστασία, κάτι το οποίο όμως δεν ισχύει. Και έχω την εντύπωση ότι δεν πιστεύουμε στις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες. Δεν λαμβάνουμε υπόψη τις αυτοαπασχολούμενες γυναίκες όπως θα έπρεπε, διότι παραμένουν στην ε, ε, αλυσίδα της επιχείρησης και βρίσκονται στην ίδια θέση με τους άντρες και υποτιμώνται. And sometimes uh, I think that uh, we και μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι δεν μας απασχολούν εξίσου οι γυναίκες αυτοαπασχολούμενες, οι οποίες είναι ε, δυνατές, είναι αρκετά δυνατές και καταβάλουν επίπονες προσπάθειες να ανταποκριθούν. Και έχουν και πολλούς εργαζόμενους στη δούλεψή τους. Αυτά ήθελα να σας πω εν ολίγης. Eh, Ευχαριστώ θερμά και ζητώ συγγνώμη που δεν είναι δυνατή η διερμηνία προς όλες τις ε, γλώσσες σε κάθε συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Φιγερέιδο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πράγματι το θέμα του γλωσσικού είναι αρκετά σημαντικό αλλά θα ήθελα να σας μιλήσω για αυτή τη γνωμοδότηση και εγώ είμαι ε, η συγγήτρια γνωμοδότηση στην Επιτροπή Βιομηχανίας και είναι ένας από τους ε, τομείς όπου τίθεται το θέμα της ισότητας. Πολύ έντονα. Γνωρίζουμε ότι η μεγάλη μισθολογική διαφορά έγκυται, βρίσκεται μάλλον στον τομέα του, της βιομηχανίας. Ε, η διαφοροποίηση αγγίζει τα όρια του 30%. Ε, στην Επιτροπή αυτή καταρτήσαμε μία, ε, μία έκθεση για το ρόλο των γυναικών στη βιομηχανία, όπου διαπιστώνουμε αυτές τις λήψεις και ανισορροπίες. Είναι ένας από τους τομείς όπου η ανεργία είναι πάρα πολύ υψηλή και οι γυναίκες αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες για να προωθήσουν ε, μία αξιοπρεπή εργασία. Συμφωνώ σε γενικές ε, γραμμές. με την παρουσίαση της συναδέλφου, η κυρία Μπρίτα Τόμσον, και νομίζω ότι ίσως θα πρέπει να μιλήσουμε και για αυτό το θέμα εμπολής και πώς οι εργαζόμενες γυναίκες στο βιομηχανικό τομέα αποτελούν αντικείμενο μεγάλων μετασχηματισμών και πολλές φορές είναι καταδικασμένες στην ανεργία. Παραμένουν δηλαδή μεγάλες ε, μισθολογικές διακρίσεις. Αυτή η πραγματικότητα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από την ε, Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Φιγερέιδο. Δίνω το λόγο στην κυρία Τόμσεν για την τελική παρέμβαση στη συζήτηση αυτή. Παρακαλώ κυρία Τόμσεν. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι πολλά βασικά ζητήματα θίγησαν και προστέθηκαν σε αυτή την έκθεση που με βρίσκουν σύμφωνοι. Νομίζω ότι θα πρέπει να φτάσουμε σε ένα στόχο 75%. Είναι ε, στόχος 25% γυναίκες στην αγορά εργασίας και θα πρέπει να έχουμε ένα σύστημα το οποίο να συνδυάζει την ιδιωτική με την επαγγελματική ζωή. Το 71% των γυναικών στη χώρα μου εργάζονται και έχουν μεγάλη ευθύνη και στο μέα του μεγαλώματος των παιδιών. Υπ' αυτή την έννοια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη αυτά τα δεδομένα, διότι χρειαζόμαστε εργατικό δυναμικό στην αγορά εργασίας ε, τη στιγμή που θα αυξηθεί ο αριθμός των ε, συνταξιοδοτηθέντων και θα βρίσκονται πολύ λιγότεροι στην αγορά εργασίας επίσης, θα πρέπει να μας απασχολήσει και ο βιομηχανικός τομέας, όπου επέρχονται πολλές αλλαγές και ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, γιατί αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ιδιαίτερα. Μιλάμε για την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπου λέμε ότι το 2020 το 20% της οικονομίας θα πρέπει να, της ενέργειας θα πρέπει να βασίζεται στις ανανεώσιμες. Σήμερα βρισκόμαστε σε ένα 9%, άρα θα πρέπει να διπλασιάσουμε και αυτό είναι το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ε, δεσμευτικό στόχο αυτό το 20%. Γι' αυτό θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας και σε αυτό το τομέα, στη μείωση του διοξίδιου του άνθρακα και στην αποδοτικότητα της ενέργειας. Ελέχθη ότι οι πολλές θέσεις, πολλές θέσεις εργασίας σε σχέση με τη μείωση εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα θα είναι εργασίες που δεν θα αφορούν χρήση υψηλών προσόντων. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, γιατί οι γυναίκες θα πρέπει να ε, μπορούν να έχουν εκπαίδευση ώστε να γίνουν ε, μηχανικοί. Διότι πολλές, πολύ λίγες γυναίκες είναι ηλεκτρολόγοι. Ξέρετε ότι στις περισσότερες χώρες πληρώνονται πάρα πολύ καλά και θα, θα χρειαστούμε πολλούς ηλεκτρολόγους που θα πρέπει να έρθουν ε, στις επιχειρήσεις, στις οικίες, για να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε εξοικονόμηση της ενέργειας για εξοικονόμηση χρημάτων, έτσι ώστε να μειώσουμε την κατανάλωση ενέργειας. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι πολύ λίγες γυναίκες βρίσκονται σε αυτό τον τομέα, απασχολούνται σε αυτό τον τομέα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Θα φύγω τώρα γιατί θα πρέπει να μιλήσω με τα ε, συνδικάτα των ε, δανών δασκάλων για να βελτιώσουμε το κείμενο. Καλή επιτυχία στην επόμενη σας συνεδρίαση κυρία Τόμσεν. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και την κυρία Τόμσεν για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής. 11 Μαΐου, 12 η ώρα, είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή 22 και 23 Ιουνίου. Η Επιτροπή Απασχόλησης θα ψηφίσει 14 Ιουλίου και... και το θέμα θα συζητηθεί στην Ολομέλεια τον Σεπτέμβριο. Επανερχόμαστε τώρα στο σημείο 4 της ημερησίας διάταξης που είναι η κοινωνική ενσωμάτωση των γυναικών που ανήκουν σε ομάδες εθνοτικών μειονοτήτων. Όπως θα θυμούνται οι συνάδελφοι, οι συντονιστές συμφώνησαν τον Νοέμβριο να εκπονηθεί έκθεση πρωτοβουλίας για το θέμα αυτό. Είχαμε και δημόσια κρόαση στις 7 Απριλίου για να ετοιμάσουμε την ε, έκθεση πρωτοβουλίας αυτή. Η συγγήτρια μας είναι η κυρία Παρβάνοβα και της δίνω το λόγο για να ε, κάνει μια εισαγωγή στην όλη συζήτηση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και όλους τους συναδέλφους γιατί ανέλαβα ένα πολιτικό πολύ ευαίσθητο ζήτημα στην εκθεσή μου και χαίρομαι πάρα πολύ που η Επιτροπή μας έχει μία συνεπή προσέγγιση από την έκθεση της κυρίας Γιαρόκα από το 2006, της κυρίας Κράτσα επίσης, για τις γυναίκες και την αμοιβή. Χρησιμοποίησα πολλές από αυτές τις πληροφορίες για την έκθεση που σας παρουσιάζω σήμερα. Η συζήτηση αυτή ακολουθεί την εξαιρετική ακρόαση που κάναμε και που μας επέτρεψε να δούμε πόσα πολλά ζητήματα υπησέρχονται. Επίσης η ακρόαση μας βοήθησε πολύ στη σύνταξη της συγκεκριμένης έκθεσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους σκιώδεις συζητητές που με βοήθησαν πάρα πολύ, όλους τους συναδέλφους. Ελπίζω να είχαν χρόνο οι συνάδελφοι να διαβάσουν ε, κυρίως την αιτιολογική έκθεση που επεξηγεί λεπτομερέστερα τι προσπάθησα να επιτύχω στην έκθεσή μου. Υπήρχαν ορισμένα ζητήματα που ετέθησαν ε, στις πρώτες συζητήσεις για την ε, εμβέλεια της έκθεσης, ε, γυναίκες μετανάστες, ε, γυναίκες εθνοτικών μειονοτήτων, γυναίκες ρομ, εξού και το πολιτικά ευαίσθητο του ζητήματος. Και ένα από τα βασικά θέματα για μένα είναι ότι η έκθεση αυτή προσπαθεί να τονίσει το εξής. Όταν μιλάμε για ισότητα των φίλων μιλάμε για όλες τις γυναίκες, αλλά στην πραγματικότητα δεν εποφελούνται όλες οι γυναίκες και δεν εποφελούνται όλες οι γυναίκες και από τις πολιτικές ένταξης. Συνεπώς, θα ήθελα να υπάρξει ένας ειδικό ορισμός, ειδικότερα για τις εθνοτικές μειονότητες ε, ή τις ιστορικές μειονότητες ή όπως θέλουμε μπορούμε να τις αποκαλέσουμε. Ο στόχος είναι που έχει σημασία και ο στόχος είναι να δούμε πώς όλες οι γυναίκες, πώς όλοι μπορούν να επωφεληθούν από τη χάρτα ε, θεμελιωδών δικαιωμάτων. Και δεδομένου ότι κατά την ακρόαση ακούσαμε ότι κάποια κράτη-μέλη δεν έχουν στατιστικά στοιχεία γιατί στην δική τους νομοθεσία δεν επιτρέπεται να συλλέγονται δεδομένα βάσει ε, εθνοτικών ε, κριτηρίων, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να το θέσω και αυτό και να ε, κάνουμε ένα επιπλέον βήμα προς τη Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων η ισότητα αφορά όλους, ανεξαρτήτως από το ιστορικό του, ανεξαρτήτως του ιστορικού του. Ε, και όσον αφορά τον τίτλο της έκθεσης θα ήθελα να τονίσω τις ε, πολλές πτυχέ. Καταρχά ε, η ένταξη, η πολιτική ένταξη, δεύτερον η ισότητα και τρίτον οι εθνοτικέ μειονότητε. Θα ήθελα να εξετάσω διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την κοινωνική ένταξη των γυναικών από εθνοτικές μειονότητες ε, με ιδιαίτερη σημασία στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στα κοινωνικά επιδόματα, στην απασχόληση, στην εκπαίδευσή τους ε, και στην οικονομική τους υποστήριξη. Προσπαθούμε να εντοπίσουμε τους τρόπους συμφιλίωσης ε, μεταξύ των διαφόρων ε, τομέων δραστηριοποίησης των τομέων αυτών ε, και να προτείνουμε νέες πολιτικές, καλύτερες πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να εξασφαλίσουμε την κοινωνική τους ε, ενσωμάτωση. Να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των γυναικών αυτών, ε, τις ανάγκες ε, ύπαρξης ίσης μεταχείρισης ε, μεταξύ όλων των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσον αφορά τις πρωτοβουλίες, τις πολιτικές, ειδικά της κοινωνικής ένταξης, ευχαρίστως εγώ να ακούσω Τροπολογίε για να βελτιώσω το κείμενό μου. Αναμένω εναγωνίω ε, την συνεργασία μου με του ε, σκιώδει εισηγητέ, προκειμένου να γίνουν πραγματικότητα όλα αυτά που προτείνουμε. Ω προ το χρονοδιάγραμμα τώρα, σήμερα θα συζητούμε την έκθεσή μου. Μέχρι τι 11 Μαου είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. 22 ε, με 23 Ιουνίου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μα και αν τα πράγματα πάνε καλά, αν δεν υπάρχουν ηφαίστεια, εκρήξει κλπ, Ελπίζουμε να ψηφίσουμε στην Ολομέλεια του Ιουλίου για την έκθεσή μου. Και θα ήθελα να προτείνω την επόμενη Δευτέρα να είναι εδώ οι συνάδελφοί μου, οι σκιώδεις, ε, οι συγητές, ε, για να κάνουμε μια προκαταρκτική συνάντηση ε, πριν ακριβώς από την καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή τροπολογιών. Στις 10 Μαΐου λοιπόν καλώ τους υπόλοιπους συναδέλφους. Θα ήθελα να ακούσω την άποψή τους γιατί είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά κυρία Περβάνοβα. Πρώτη ομιλήτρια, κυρία Μπόσκουιτ. Ehm, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την κυρία Παρβάνοβα για την ε, έκθεσή της. Αναφέρει πολλά σημαντικά σημεία και υπάρχουν ορισμένα τα οποία θα θέλω να τονίσω κι εγώ. Καταρχάς, Κάτι που νομίζω ότι απουσιάζει, και θα ήθελα να υποβάλω και τροπολογία γι' αυτό, ο ρόλος της κοινότητας, πώς ε, οι ενώσεις ε, δικαιωμάτων των γυναικών, ε, οι οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών που εκπροσωπούν τις γυναίκες αυτές, πώς τις εκπροσωπούν. Πρέπει οπωσδήποτε να συνεργαστούμε με τις οργανώσεις αυτές και, αυτές και πρέπει να ενθαρρύνουμε τις γυναίκες να είναι πιο δραστήριες σε ζητήματα όσον αφορά την εκπαίδευση, για παράδειγμα, ώστε όταν υπάρχουν διάφορες διευκολύνσεις όπως μαθήματα γλώσσας κλπ, όταν βλέπουν δηλαδή ότι υπάρχουν κάποιοι, κάποιες ε, προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση, τότε και οι γυναίκες εκείνες ε, θα ε, προσεγγίσουν τις προσπάθειες αυτές και θα προσπαθήσουν να τις αξιοποιήσουν. Και είναι κάτι το οποίο βέβαια θα έχει ως αποτέλεσμα και την καλύτερη ένταξη των παιδιών. Νομίζω λοιπόν ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αναφέρουμε δεν βοηθούμε μόνο τις γυναίκες εν βοηθούμε ολόκληρη την κοινότητα και τα παιδιά των γυναικών αυτών. Και θα ήθελα να τονίσω και το θέμα των καλών στοιχείων, των καλών δεδομένων που το έχει αναφέρει η κυρία Παρβάνοβα στην ε, έκθεσή της. Πρέπει επίσης να γνωρίζουν όλοι τα δικαιώματά τους οι εθνοδικές μειονότητες. Πολλές ε, εθνοτικές ε, μειονότητες έχουν πολλά δικαιώματα τα οποία όμως δεν γνωρίζουν. Θα ήθελα επίσης να τονίσω όταν υπάρχει πόλωση σε μια κοινωνία, για παράδειγμα η κατάσταση των Ρώμ σε, πολλές, ε, σε πολλά κράτη-μέλη, υπάρχουν και πολλές διακρίσεις, ακόμη και στα λόγια πολλές φορές. Κάτι το οποίο καθιστά ακόμη δυσκολότερη την κοινωνική ένταξη των ε, ε, γυναικών. Και το ίδιο ισχύει για τις ε, μουσουλμάνες. Για παράδειγμα, στη δική μου χώρα, τις κάτω υπάρχει ιδιαίτερη πόλωση όσον αφορά την ένταξη των μουσουλμάνων και βλέπουμε, ας πούμε, γυναίκες με μαντήλες που έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα να ε, συμμετέχουν σε προγράμματα, για παράδειγμα, άσκησης, σε διάφορες επιχειρήσεις, σε προγράμματα μαθητείας. Όλα αυτά, λοιπόν, είναι στοιχεία τα οποία πρέπει να συμπεριληφθούν στην έκθεση για να υπάρχει μία πλήρης εικόνα της κατάστασης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπόσκο. Το λόγο έχει η κυρία Μπάουερ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να επενέσω την προσέγγιση της εισηγήτριας για το θέμα αυτό, διότι είναι πολύ ευαίσθητο θέμα, πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολο θέμα. Έχω κάποιες ερωτήσεις και κάποιες παρατηρήσεις. Στο εκτιμώντας, ε, το ελέγξα σε δύο γλώσσες και ακόμα δεν καταλαβαίνω, διότι έχω την αίσθηση ότι πρόκειται για κάποιο λάθος Μιλάμε για το εκτιμώντας ΙΓ και αναφέρεται το δικαίωμα της ακαιρεότητα. Μάλλον πρόκειται για το δικαίωμα ενσωμάτωσης, ένταξης. Αν είναι όντω σωστό το κείμενο που έχω μπροστά μου, θα ήθελα κάποιες εξηγήσεις, διότι άλλο η ακαιρεότητα, άλλο η ένταξη. όσον αφορά το σημείο 4. όπου αναφέρεται η ενθάρρυνση των διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πώς μπορεί η Κομισιόν να ενθαρρύνει την ύπαρξη αυτών των διαπολιτισμικών διαμεσολαβητών. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Θα ήθελα δηλαδή διευκρινήσεις σχετικές και θα ήθελα να προσθέσω ότι σε κάποια σημεία έχω την αίσθηση ότι το κείμενο αυτό είναι ακόμα πιο αποδυναμωμένο από την ισχύουσα νομοθεσία. που προϋποθέτει την ύπαρξη θετικών δράσεων για την αντιμετώπιση της κατάστασης για την αντιμετώπιση καταστάσεων που μπορούν να θεωρηθούν διακρίσεις. με την εφαρμογή της αρχής του πολίτη, δηλαδή Μιλάμε για περιπτώσεις έμεσης διάκρισης. Πρόκειται για πολύ ισχυρό μέσο που υπάρχει στις δύο οδηγίες που έχουμε για την καταπολέμηση των διακρίσεων. Όσον αφορά το όλο θέμα, έχω την εντύπωση ότι το μπέρδεμα των παραδοσιακών μειονοτήτων με τους μετανάστες δεν είναι πολύ καλός τρόπος αντιμετώπισης. Τελικά, μπορεί να δημιουργηθεί σύγχυση. Για παράδειγμα, στο σημείο 5 μιλάμε για χρήση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξη, το οποίο όμω δεν έχει, να κάνει καθόλου με τι εθνοτικέ μειονότητε. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξη, ε, στόχο έχει την ένταξη των μεταναστών. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι απαραίτητο να γίνει σαφής διάκριση ανάμεσα στις εθνοτικέ μειονότητες που επί αιώνες ζουν στις κοινωνίες μας, να υπάρξει διάκριση αυτών από τη μία και από την άλλη των μεταναστών, των οποίων οι συνθήκες διαβίωσης και οι ανάγκες είναι τελείως διαφορετικές. Με την προϋπόθεση αυτή, να μην γίνεται δηλαδή διάκριση ανάμεσα σε δύο τελείως διαφορετικές ομάδες, έχω την εντύπωση ότι θα χάσει σε αξία η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Κίλ Νίλσεν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Να ευχαριστήσω την κυρία Παρβάνοβα γιατί ανέλαβε ένα θέμα πάρα πολύ δύσκολο και χρειάζεται πολύ θάρρος και κουράγιο, οπότε την ευχαριστώ. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Θα το ξαναπώ δυστυχώς. Υπάρχει... είναι μάλλον ε, δύσκολο να συζητήσουμε έτσι γενικό στο θέμα των εθνοτικών μειονοτήτων, ε, τους μετανάστες που μπορεί να είναι νόμιμοι ή παράνομοι και υπάρχουν επίσης και οι ετώντες, ε, οι άσυλο. Οπότε πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ αυτών των ομάδων. Δεν είναι δυνατόν να τις συζητούμε όλες μαζί γιατί τα προβλήματα δεν είναι τα ίδια, τα αιτήματα δεν είναι τα ίδια και τα μέτρα, τα μέσα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε δεν είναι υποχρεωτικά ίδια. Οπότε νομίζω ότι πρέπει να είναι σαφέστερη η διάκριση μεταξύ των ε, κατηγοριών αυτών. Το θέμα τώρα του ακαιρεότητα ή ενσωμάτωση, εντεγκριτέ ή ε, εντεγκρασιόν στο γαλλικό κείμενο, αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το διευκρινίσουμε απλώς γλωσσικά. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Παλιαδέλη. Παρακαλώ. Εκτός μικροφώνου δεν ακούγεστε. να ευχαριστήσω την κυρία Παρβάνοβα για το θάρρος να αναλάβει ένα τέτοιο δύσκολο αλλά τόσο σημαντικό θέμα. Να δηλώσω ότι δεν πρόλαβα να το μελετήσω παρά μόνο από την Παρασκευή μεσημέρι που είχα τη δυνατότητα να το έχω στα χέρια μου ε, και να συμφωνήσω με τις ε, κυρίες που μίλησαν πριν από μένα ότι πραγματικά ε, υπάρχει ένα ζήτημα μιας μικρής ασάφειας ανάμεσα, μιας ασάφειας ανάμεσα στην, στους όρους μειονότητες, εθνικές, εθνοτικές μειονότητες και ε, μετανάστες. Αυτό νομίζω ότι θα έπρεπε να αποσαφινιστεί ε, όταν μάλιστα ε, ούτε καν η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει καταλήξει σε ε, σαφείς ορισμούς των, εθνικών, εθνοτικών μειονοτήτων έχει αποφύγει και φαίνεται πολύ καλά στην έκθεση της κυρίας Παρβάνοβας το ε, ε, αυτή η δυσκολία θα έλεγα ότι θα ήταν ίσως πιο περισσότερος ασφαλές να μην εμπλακεί στην έκθεση το ζήτημα της, του ορισμού των μειονοτήτων εθνοτικών ή άλλων και να αντιμετωπιστούν το σύνολο των γυναικών που δεν έχουν τα τυπικά δικαιώματα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θεωρητικά οι γυναίκες των μειονοτήτων που ζουν και έχουν τα νομικά, ίσα νομικά δικαιώματα με τις υπόλοιπες γυναίκες που δεν ανοίγουν σε μειονότητες, τυπικά ε, δεν διαφέρουν από εκείνες. Αντίθετα, θα έλεγα ότι συχνά προβλήματα προκύπτουν στις γυναίκες αυτές από τις δικές τους, από τους χώρους στους οποίους ε, εντάσσονται. Δηλαδή η πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν είναι αναγκαστικά ε, ε, μια απόφαση που την παίρνει μόνη της μια γυναίκα μιας εθνικής μειονότητας, συχνά της επιβάλλεται από το δικό της περιβάλλον, από, τα δικά της, από τις δικές της αναστολές. Επομένως, καμιά φορά δεν φταίει το κράτος μέλος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση, καμιά φορά φταίει το περιβάλλον από το, στο οποίο εντάσσεται εθνοτικά. Επομένως, ένα μέρος κάπου πρέπει να, να, διατυπωθεί και αυτό το ε, ζήτημα, εκτιμώ. Ε, επειδή συμβαίνει να είμαι ε, shadow reporter στην ε, έκθεση, σίγουρα θα κουβεντιάσουμε περισσότερο για τέτοια ζητήματα, αλλά θα ήθελα να γυρίσω στην βασική μου αντίρρηση σε αυτή την πολύ σοβαρή προσέγγιση για ε, ένα πολύ, σημαντικό θέμα, ότι από τη στιγμή που δεν έχουμε ορισμούς από την, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είναι, ίσως θα ήταν σκοπιμότερο να μην επανα να μην ζητήσουμε να τους ορίσουμε εμείς εδώ σε αυτή την Επιτροπή. Εκτιμώ ότι αυτή η έκθεση πρωτοβουλίας θα αποκτήσει μεγαλύτερη αξία, παραπέμποντας την κυρία Μπάουερ, αν αποφύγουμε τον σκόπελο που ε, ε, προκύπτει από το τι είναι ε, εθνοτική μειονότητα, τι είναι migrants κλπ. Επομένως, εμείς οι δυο θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα ακούσουμε τώρα τη θέση της Επιτροπής. Η κυρία Χέιτειλ, παρακαλώ. Καλησπέρα. Εγώ είμαι από το τμήμα ισότητας ε, των φίλων ε, ε, της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το σχέδιο ε, έκθεσής της και όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοί σας πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα η, η ένταξη των γυναικών των, εθνικών, των εθνοτικών μειονοτήτων και πολλές φορές ε, βλέπουμε ότι είναι αντικείμενο διάκρισης και γι' αυτό ακριβώς ε, ο δικός χάρτης 2006-2010 ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ισότητα των φύλων ασχολείται ειδικότερα με το θέμα αυτό και αποτελεί θέμα προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι γεγονός τώρα ότι η κατάσταση αυτή των γυναικών γυναικών αυτών ε, χρειάζεται κινητοποίηση πολλών πολιτικών, όχι μόνο ισότητα των φύλων ε, και κατά των διακρίσεων, αλλά και στο πλαίσιο της ε, απασχόλησης και πολλών άλλων τομέων που υπησέρχονται και τους οποίους αναφέρει η έκθεση. Ενδεχομένως να υπάρχουν ορισμένα ζητήματα συγκεκριμένα επί των οποίων θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή το γεγονός ότι συχνά μιλάμε για τις πολιτικές ένταξης και συχνά καταλαβαίνουμε ότι αφορούν ε, γυναίκες τρίτων χωρών, ε, μετανάστριες δηλαδή, και μιλούμε για το πώς θα ενταχθούν καλύτερα στη χώρα που τις φιλοξενεί. Όμως ε, μιλάμε κυρίως για την κοινωνική ένταξή τους και εννοούμε κυρίως την κοινωνική τους ένταξη σε όλα τα κοινωνικά προγράμματα και με όλες τις συνέπειες που μπορεί να έχει αυτό. Και δεν μιλάμε μόνο για γυναίκες τρίτων χωρών. Άρα λοιπόν η ενσωμάτωση και άλλο η ένταξη. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Η κοινωνική ένταξη με αυτήν την έννοια δηλαδή. Όσον αφορά τη συλλογή των ε, δεδομένων όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως είναι κάτι το πάρα πολύ δύσκολο. Η ανάπτυξη της συλλογής των δεδομένων ε, ανά εθνοτική μειονότητα είναι πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί μερικά κράτη-μέλη δεν το επιτρέπουν στην ομοθεσία του. Βεβαίω, υπάρχουν κάποιοι τρόποι που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διάφορες στατιστικές μεθόδους για να συμπεριλάβουμε, ε, για να ε, συλλέξουμε τα στοιχεία αυτά όπως για παράδειγμα την ε, υπηκότητα, τα χρόνια διαμονής σε μια χώρα ε, ή την ε, χώρα γέννησης του ατόμου και πολλές φορές υπάρχουν και μητρώα ενσωμάτωσης των μεταναστών και των απογόνων τους που συνδυάζονται για παράδειγμα με, το, με, το, τη χώρα γέννησης των μεταναστών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να προωθήσει τη χρήση τέτοιου είδους μεθόδων ώστε να μπορέσουμε ε, από το 2014 να έχουμε καλύτερα στοιχεία στη διάθεσή μας από όλα τα κράτη-μέλη. Κάτι ακόμη θα ήθελα να πω σε σχέση με την εκπαίδευση. Η Περιεκτική εκπαίδευση είναι αυτή που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βελτίωση δηλαδή της πρόσβασης ε, σε συγκεκριμένα είδη εκπαίδευσης για συγκεκριμένες ε, εθνοτικές μειονότητες. Όμως είναι γεγονός ότι πολλές φορές τέτοιου είδους ομάδες βρίσκονται σε ε, πλαίσιο χαμηλότερης εκπαίδευσης και εδώ υπάρχει δηλαδή ένα χάσμα Προσπαθούμε λοιπόν να βελτιώσουμε την πρόσφαση σε ποιοτική εκπαίδευση με συγκεκριμένη υποστήριξη των συγκεκριμένων ομάδων, είτε με μεγαλύτερα, με περισσότερο στοχευμένα προγράμματα, είτε με άλλους τρόπους. Κάτι άλλο το οποίο επίσης αναφέρατε κι εσείς, ε, η ευαισθητοποίηση των ε, νομικών και νομομαθών για τον τομέα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη αναλάβει προγράμματα κατάρτισης ε, για νομικούς και νομομαθείς ε, στο πλαίσιο της ισότητας των φύλων και της νομοθεσίας ε, κατά των διακρίσεων και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό πιστεύουμε ότι θα έχει πολλά, πολύ σημαντικά αποτελέσματα γιατί πολλές φορές οι νομικοί δεν γνωρίζουν την ευρωπαϊκή νομοθεσία που, υπάρχουν, που υπάρχει για τα ζητήματα αυτά. Όσον αφορά τώρα το θέμα της, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας ε, των ε, Φύλων, γνωρίζετε ότι τώρα ιδρύεται και θα καταστεί ανεξάρτητο και λειτουργικό από τον ε, Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Θα συλλέγει δεδομένα και θα... Ε, ε, γνωστοποιεί δεδομένα σχετικά με το θέμα και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό Ίσως θα έπρεπε να αναφέρεται μάλιστα και στην έκθεση. Κάτι τελευταίο που θα ήθελα να πω, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, έχουμε μία έκθεση εμπειρογνωμόνων για τις εθνοτικές μειονότητες και τις γυναίκες ΡΟΜ που ε, αναφέρει στοιχεία από 13 ευρωπαϊκές χώρες και περιγράφει το πρόβλημα του ορισμού των εθνοτικών μειονοτήτων ή των μειονοτήτων καθαρά και εξετάζει επίσης την κατάσταση των γυναικών εθνοτικών μειονοτήτων ε, στην πρόσβαση στην ε, ιατροφαρμακευτική ε, περίθαλψη, στην υγεία, στην ε, απασχόληση, στην εκπαίδευση και σε άλλους τομείς και νομίζω ότι και αυτό θα μπορούσε να βοηθήσει ως στοιχείο στην σύνταξη της έκθεσης. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ θερμά η κυρία Παρφάνοβα Έχει το λόγο για την τελική παρέμβαση. Παρακαλώ. Ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους που μου δώσαν, ε, μάλλον σχολίασαν την πρότασή μου και βεβαίως Μιλάμε για τις εθνικές μειονότητες και τους μετανάστες, γι' αυτό αναφέρθηκα ειδικά σε αυτό και είπα ότι αν θέλουμε να μπούμε σε έναν ορισμό, είμαστε τόσο φιλόδοξοι, βεβαίως αναγνωρίζουμε ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ εθνικών μειονοτήτων και τους μετανάστες γενικότερα, όχι ειδικά για τις γυναίκες, αλλά και για τις γυναίκες. Τότε θα αντιμετωπίσουμε εθνικά και πολιτικά προσκόμματα. Δεν θα ήθελα να εξανεμιστεί αυτή η έκθεση στον διάλογο μεταξύ Κομισιών Συμβουλίου, Κοινοβουλίου, Κρατών Μελών και πολιτικών ομάδων. Για μένα δεν έχει τόσο σημασία πώς ε, οι γυναίκες αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας, εκπαίδευσης, ε, προβλήματα στο σεξουαλικό τομέα. Αυτό που έχει σημασία είναι το πώς αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα σε εθνικό επίπεδο, σε επίπεδο πολιτικής, αλλά όχι σε αυτή την έκθεση, διότι υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν διαφορετική προσέγγιση για να δούμε κατά πόσο μια ομάδα είναι μια εθνοτική μειονότητα, ε, εάν πρόκειται για ετούντες άσυλο, για μετανάστες και ούτω καθεξής. Ορισμένες μη κυβερνητικέ κατά την ακρόαση μίλησαν για μετανάστες τρίτης γενεάς και έθεσαν το ζήτημα κατά πόσο θεωρούνται εθνική μειονότητα ε, ή αν έχουν πια εγκατασταθεί για τα καλά. Γιατί πολλές φορές μιλάμε και για το Ισλάμ. Στο Βέλγιο ή στην Ελλάδα, όπως είπε η συνάδελφος, υπάρχει διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με την ιστορική εγκατάσταση αυτής της μειονότητας και εδώ στο Βέλγιο οι Φλαμανδοί και οι Βαλόνοι δεν μπορούν να θεωρήσουν ορισμένες κατηγορίες ως μειονότητα ή μη. Γι' αυτό δεν πρέπει να υπάρξει παρανόηση. θα ήθελα να εστιάσουμε την προσοχή μας στα προβλήματα, στην έκβαση και τον αντίκτυπο των πολιτικών που προβάλλουμε. Για να ενισχύσουμε την προσέγγιση μας για την επίλυση αυτών των προβλημάτων. Σε σχέση τώρα ο, ορισμένες προτάσεις, σας ευχαριστώ που μιλήσατε για τις μη κυβερνητικέ, για την ε, ε, εκπαίδευση, Έχουμε ένα χρονικό περιορισμό για αυτή την ε, έκθεση. Έχουμε ανοιχτή προσέγγιση. Σίγουρα υπάρχει χώρος για τροπολογίες και μπορώ να δεχτώ όλες αυτές τις προτάσεις ως προς τη συλλογή δεδομένων. Συμφωνώ με την Επιτροπή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να συλλέγουμε στοιχεία μόνο για λόγους απασχόλησης. Γιατί αν μιλάμε για ιστορικές ε, μειονότητες, για την χώρα προέλευσης ή χώρα γέννησης, όλα αυτά δεν έχουν και τόσο μεγάλη σημασία. Θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να κοιτάξουμε πέρα από τη συλλογή δεδομένων ως προς τη, τους οργανισμούς για την ισότητα των δύο φύλων, ίσως είναι γλωσσικό το θέμα. Συμφωνώ ότι η λέξη implementing δεν είναι η σωστή. Ήθελα να πω ότι οι προτάσεις μας, για τα, οι προτάσεις μας αφορούν τα κατάλληλα μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν. Και θα πρέπει να γίνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης έτσι ώστε να συμμετέχουν οι κοινότητες, αλλά βασίζομαι στις τροπολογίες και τις προτάσεις των συναδέλφων και νομίζω ότι θα βρούμε έναν τρόπο να ε, περάσει αυτό το ε, θέμα θετικά και να έχουμε και την κατάλληλη υποστήριξη. Γιατί αν είναι κάτι που το αφήσουμε να πεθάνει από φυσικό θάνατο, τότε δεν θα είμαστε συνεκτικοί στην ε, προσέγγιση μας. Θα πρέπει να φτάσουμε μέχρι τέλους σε αυτή την πορεία και στόχος μας είναι να βρούμε ε, μία λύση σε ένα ζωτικό ζήτημα το οποίο δεν μπορούσαμε να αποφύγουμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Παρβάνοβα. Ήδη αναφερθήκατε στο χρονοδιάγραμμα. Για το θέμα αυτό μπορούμε λοιπόν να προχωρήσουμε στο σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης που είναι η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Είναι η λεγόμενη Υπηρεσία Εξωτερικών Υποθέσεων. Τον Μάρτιο η Επιτροπή μας αποφάσισε να εκπονήσει γνωμοδότηση για το θέμα αυτό που έχει να κάνει με διάφορα μέτρα που σχετίζονται με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Τα αρχικά είναι EEAS. Σήμερα θα συζητήσουμε την δημιουργία Τη Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξεταρικής δράση. Άλλε πτυχέ έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότηση, τον προπολογισμό δηλαδή, το προσωπικό κλπ. Η γνωμοδότηση που έχουμε σήμερα υπάρχει μόνο στα αγγλικά. Αλλά πριν το τέλος της προθεσμίας για την υποβολή τροπολογιών θα υπάρχει το κείμενο σε όλες τις γλώσσες. Η κυρία Φρανσίσκα Μπραντνερ είναι αρμόδια από την Επιτροπή μας. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να παρευρεθεί εδώ σήμερα. Η κυρία Κορνέλισεν αντικαθιστά την κυρία Μπραντνερ. Της δίνω λοιπόν το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Μπραντνερ έπρεπε να ε, φύγει, να αποχωρήσει, διότι θα γεννήσει σε δύο εβδομάδες, θα επανέλθει το Σεπτέμβριο. Έχει εργαστεί πολύ σκληρά για την έκθεση αυτή. Ήταν συντονίστρια, μία από τους ε, συντονιστές της ΑΦΕΤ και εργάστηκε για την συγκρότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Θα αναλάβω εγώ αυτό το έργο με τον Ερίκα Λούνατσεκ που ήταν ε, ε, από κοινού συντονίστρια με την ε, Κατερίνα Μπραντνερ και ξέρει για την δράση αυτής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας. Χαίρομαι διότι και η δική μας Επιτροπή γνωμοδότησε για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικές Δράσεις. Υπάρχουν πολλές, πολλοί φορείς των οποίων η σύσταση γίνεται χωρίς να ληφθεί η υπόψη διάσταση ισότητας των δύο φύλων και το mainstreaming αυτό είναι ε, πολύ δύσκολο να γίνει εκ των υστέρων όταν όλα έχουν παγιωθεί είναι πολύ δύσκολο να ενσωματωθεί η διάσταση της ισότητας των δύο φύλων. Άρα, εδώ μπορούμε εξ αρχής να ενσωματώσουμε την ισότητα των δύο φύλων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Ε, αναφερθήκατε και σε μερικά σημεία που αφορούν την ισότητα του προσωπικού και ως προς το mainstreaming για το περιεχόμενο. Μιλάμε για ένα 50-50 μια κατανομή 50-50 σε επίπεδο αρχηγών αντιπροσωπιών αλλά και σε όλα τα άλλα επίπεδα του προσωπικού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όχι μόνο γιατί χρειαζόμαστε το input των γυναικών στις εξωτερικές μας πολιτικές, αλλά γιατί θα πρέπει να ορίσουμε ε, μια παραδειγματική σχέση. Δύο μήνες πριν βρέθηκα στη Βοσνία και μίλησα με ορισμένες γυναικείες οργανώσεις όπου μου είπαν ότι ακούν πολλά λόγια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το πόσο είναι σημαντικό να κατέχουν οι γυναίκες θέσεις σημαντικές, αλλά δεν είδαν ποτέ γυναίκες σε υψηλές θέσεις ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση που να μεταβεί σε εκείνες. Και αυτό αποτελεί πολύ κακό παράδειγμα. Θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε το σωστό παράδειγμα προς τα έξω. Και θα ήθελα να τονίσω ότι θα πρέπει να έχουμε ένα αρκετά υψηλό ποσοστό γυναικών σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να μην παγιωθούν αρνητικές καταστάσεις. Υπάρχουν πολλές διεθνείς οργανώσεις που ε, προβάλλουν παχιά λόγια για την ισότητα των δύο φίλων, αλλά δυστυχώς ε, βλέπουμε ότι δίνεται πολύ αρνητικό παράδειγμα. Γι' αυτό προτείνουμε να ε, συσταθεί ένα τμήμα που να ενσωματώσει την ισότητα των ε, δύο φίλων στην εξωτερική δράση. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, στην Αϊτή μετά το σεισμό στους καταβλισμούς προσφύγων ξέρουμε ότι θα πρέπει να προσδώσουμε μεγάλη σημασία στη διάσταση των φύλων γιατί διαφορετικά υπάρχει ε, υψηλός, υψηλοί δείκτες ε, βιασμών στους καταβλισμούς. Χρειαζόμαστε ένα τμήμα στην υπηρεσία εξωτερικής δράσης για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο. Γιατί ακόμα ε, και το θέμα της υγιεινής, δηλαδή διαφορετικές τουαλέτες για άνδρες και γυναίκες, έχουν μεγάλη σημασία στους ε, καταβλισμούς αυτούς. Επίσης θα έπρεπε να έχουμε κατάρτιση του διπλωματικού προσωπικού έτσι ώστε ε, εκείνοι που βρίσκονται επί να είναι ευαισθητοποιημένοι στο θέμα αυτό. Επίσης, ε, δεν θα πρέπει ο προπολογισμό να είναι ένας χάρτινος ε, τίγρης και να έχουμε μία αποτίμηση για την πραγματική ισότητα, έτσι ώστε δημοκρατικά να μπορέσουμε να ελέγξουμε την υπηρεσία εξωτερικής δράσης για να ξέρουμε τι κάνει και η ύπατη εκπρόσωπος. Ελπίζω ε, οι άλλες ομάδες να μπορέσουν να με υποστηρίξουν. Ehm, Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Αντιπρόεδρο Μωρέν είναι η πρώτη ομιλήτρια. Euh, Σα ευχαριστώ πολύ. Η, η παρέμβασή μου ε, σχετίζεται με τη θέση της Μαρία Ναντέλτσεβα που είναι σκιώδης για το ΕΛΚ ως προς το, ε, την γνωμοδότηση Μπράντνερ για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης. Η κυρία Ντέλτσεβα αυτή τη στιγμή ε, λείπει, βρίσκεται αλλού και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στη σημερινή συζήτηση. Μου ζήτησε λοιπόν να την εκπροσωπήσω και υπ' αυτή την ιδιότητα ε, μιλώ δηλαδή, εκφράζω τη δική της, εκφέρω τη δική της άποψη. Θα ήθελα να χαιρετήσω το προσχέδιο ε, αυτό της κυρίας Μπραντνερ ως προς την πρόταση του Συμβουλίου για τη σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Εάν η Επιτροπή ε, των Δικαιωμάτων των Γυναικών και της ισότητας των γυναικών ε, μπόρεσε και θα μπορέσει να συντάξει ε, μία γνωμοδότηση, αυτό σημαίνει ότι λαμβάνουμε υπόψη την ισότητα που κατέχει πρώτη τη σημασία στην ε, σύσταση αυτής της υπηρεσίας. Αυτή η γνωμοδότηση θέλει να εξεύρει λύση στην ανισορροπία και μη ισότητα των δύο φύλων εάν δεν θέσουμε επί χάρτου τους στόχους μας επί του θέματος. Η σύσταση αυτής της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης θα πρέπει να επαυξήσει την την ορατότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανά τον κόσμο. Η υπηρεσία αυτή επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να διαθέτει μία διάρθρωση η οποία να έχει ειδικό βάρος στο διεθνές προσκήνιο έτσι ώστε να ενδυναμώσουμε την δυνατότητα δράσης μας σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει λοιπόν αυτή η βιτρίνα της Ευρώπης να μπορέσει με τις αντιπροσωπείες της να βρίσκεται σε όλα τα σημεία του κόσμου αλλά με βάση την ισορροπία εκπροσώπησης ανδρών και γυναικών. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου είναι δύσκολες. Τα κράτη-μέλη δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν με το Κοινοβούλιο επιθεμάτων ελέγχου του προϋπολογισμού ως προς την ε, διάφραση αυτής της υπηρεσία υπό την αιγίδα της Κάθριν Άστον. Η ισότητα ανδρών γυναικών είναι ύψης της σημασίας και θεωρώ ότι δεν πρέπει να επιβαρύνουμε τη συγγραφή υποχρεώσεων των διαπραγματεύσεων τη στιγμή που μιλάμε για συγκεκριμένες αρμοδιότητες και επιμερισμό τους. Η κυρία Άστον θα διορίσει του, τα πρόσωπα με τα κατάλληλα προσόντα που αφορούν και άνδρες και γυναίκες και επ' αυτής της αρχής θα πρέπει να βασιστούμε έτσι ώστε να έχουμε μία σωστή διπλωματική εκπροσώπηση. Ευχαριστώ. Υπάρχει άλλος που θέλει να πάρει το... Om Εάν όχι, να ρωτήσω την κυρία Κορνέλησεν αν θέλει να κάνει κάποια ε, τελική παρέμβαση. Παρακαλώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Μωρέ εκ μέρους της κυρίας Μπραντνερ για τις παρατηρήσεις της. Γνωρίζω ότι είναι δύσκολες οι διαπραγματεύσεις και ότι σαφώς θα πρέπει ως Επιτροπή Γυναικών να προβάλλουμε τις θέσεις μας. Δεν νομίζω ότι κάτι τέτοιο θα περιπλέξει τα πράγματα. Υπάρχουν, πράγματα πολύ, υπάρχουν θέματα πολύ πιο καυτά από αυτό. Είμαι ευγνώμων για την υποστήριξή σας. Θα περιμένω να δω τι επικοδομητικές ε, τροπολογίες θα υποβληθούν. Ευχαριστώ. Το χρονοδιάγραμμα έχει ως εξής. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών 8 Μαΐου στις 12 η ώρα. Θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή στις 22 και 23 Ιουνίου. Προχωράμε. Στο θέμα υπαριθμών 7 της ημερησίας διάταξης είναι το τελευταίο σημείο της ημερησίας διάταξης για σήμερα διότι έχουμε στις 5 ε, και 4 την κοινή, την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Τώρα θα συζητήσουμε την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Οι συντονιστές της Επιτροπής μας ε, ε, αποφάσισαν τον Σεπτέμβριο, συμφώνησαν μεταξύ τους, σχετικά θέματα που θα διαλευκάνουν πώς εφαρμόζουν τα διάφορα κράτη-μέλη την, την ε, νομοθεσία περί ισότητας. Έδωσαν εντολή στην Πρόεδρο να εκπονήσει προτάσεις ε, σχετικά με το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Σήμερα λοιπόν περιμένουμε μια γενική παρουσίαση από εκπρόσωπο της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων. Πρόκειται για ένα πρώτο βήμα μετά τη συζήτηση που είχαμε μεταξύ των συντονιστών. Καλωσορίζω λοιπόν από την Κομισιόν, από τη Γενική Διεύθυνση για την Απασχόληση, τον κύριο Φερνάντο Μπορένα που θα μας κάνει μια γενική παρουσίαση. Παρακαλώ. Περιμένουμε να λάβουμε τις πληροφορίες που έχετε να μας δώσετε. Παρακαλώ. Merci, Madame la Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ που προσκαλέσατε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να παρουσιάσει ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα της καθημερινής της εργασίας ε, που συχνά υποτιμάται εκτός ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και είναι λιγότερο αισθητή και ορατή από άλλα νομοθετικά ζητήματα. Θα κάνω μια γενική παρουσίαση όπως είπατε κι εσείς και θα ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η κοινοτική νομοθεσία όσον αφορά τα φύλλα ουσιαστικά έγινε από το 2002 μέχρι το 2010. Το 2002 έγινε μια πρώτη σοβαρή αλλαγή της πρώτης οδηγίας. Το 2004 είχαμε μια οδηγία που για πρώτη φορά επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής της ισότητας των φύλων ε, πέρα από την απασχόληση. Μετά το 2006 μια αναδιατύπωση που αφορούσε 7 οδηγίες ε, και τέλος, ε, παρά το γεγονός ότι δεν θα ασχοληθώ με αυτήν σήμερα, μία οδηγία που μόλις εγκρίθηκε το 2010 και που εξυγχρονίζει ε, την ε, οδηγία ε, του 96 για τις ε, γονεϊκές άδειες. Θα ήθελα λοιπόν να μιλήσω για την εφαρμογή των οδηγιών αυτών, τις οδηγίες του 2004, του 2004 και του, του 2002, του 2004 και του 2006. Αυτές οι τρεις οδηγίες έχουν προθεσμίες μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο από 2000, το 2005 για την πρώτη οδηγία μέχρι το 2009 για την τελευταία οδηγία από αυτές που θα μας απασχολήσουν σήμερα. Πρόκειται λοιπόν ε, για ζητήματα που είναι αρκετά πρόσφατα και στην πρώτη φάση η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως πάντα ήταν ε, ότι έγινε όντως μεταφορά της οδηγίας ε, στις εθνικές νομοθεσίες ε, και για την πρώτη αυτή, αυτή, αυτή πτυχή της εργασίας του ελέγχου της εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας για το θέμα λοιπόν αυτό της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο και, το, της κοινοποίηση των σχετικών μέτρων από τα κράτη-μέλη η κατάσταση έχει ως εξής. Όσον αφορά την πρώτη οδηγία, την οδηγία του 2002-73, ε, όλα τα κράτη-μέλη, χωρίς καμία εξαίρεση, έχουν μεταφέρει τώρα την οδηγία αυτή ε, στο εθνικό τους ε, δίκαιο, δηλαδή έχουν αναλάβει μέτρα, δεν μιλάω ακόμη για, τα, για την ποιότητα της μεταφοράς αυτής. Όσον αφορά τώρα την οδηγία 2004 για την πρόσβαση στα αγαθά και τις υπηρεσίες, μεταφέρθηκε σε όλα τα κράτη-μέλη με την εξαίρεση εξαίρεση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Πολωνίας. Το Ηνωμένο Βασίλειο Άλλωστε, μόλις καταδικάστηκε από το δικαστήριο, γιατί μόλις διαπιστώθηκε η παράληψη του κράτους μέλους αυτού και ε, βέβαια θα ξεκινήσει η διαδικασία του άρθρου 260 που μπορεί να οδηγεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιβάλλει πρόστιμο εάν εντωμεταξύ το κράτος μέλος δεν αναλάβει τα μέτρα που χρειάζεται. Όσον αφορά την Πολωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ενημέρωσε το κράτος μέλος ότι, δεν θα, ότι έπρεπε να ε, ε, αναλάβει την ε, μεταφορά της οδηγίας και κατά πάσα πιθανότητα αυτό θα γίνει. Όσον αφορά το 2006, της ε, αναδιατύπωσης ε, δηλαδή, με προθεσμία στο 2009. Είναι λίγο πιο αρνητικά τα πράγματα. Βέβαια, τα περισσότερα κράτη-μέλη την έχουν μεταφέρει. Μόνο πέντε δεν το έχουν κάνει ή δεν έχουν πλήρως ενημερώσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα μέτρα μεταφοράς. Αυστρία, Βέλγιο, Ιταλία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο είναι τα κράτη-μέλη. Όλα αυτά τα κράτη-μέλη έχουν ε, λάβει ε, σχετική ενημέρωση που ξέρετε ότι είναι η τελευταία ε, διαδικασία πριν από τις νομικές διαδικασίες που είναι να η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, για κάποια κράτη-μέλη εξακολουθεί να ισχύει ακόμη προθεσμία απάντησης, ε, αλλά μόλις εκπνεύσει η προθεσμία αυτή, μπορεί να προσφύγει στη δικαιοσύνη αν μέχρι τον επόμενο μήνα δεν έχουμε περαιτέρω στοιχεία από τα 5-7 κράτη-μέλη που ανέφερα. Όσον αφορά τώρα την ε, ε, κοινοποίηση πρέπει να πω ότι στα κράτη-μέλη που έχουν μεταφέρει όλες τις οδηγίες είναι αρκετά πολλά, είναι αρκετά, μόνο πέντε κράτη-μέλη παραμένουν ε, για την ε, τελευταία οδηγία και δύο για το 2004. Θα ήθελα κυρία Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε, να πω το εξής, ότι με τη δέουσα επιμέλεια ασχολήθηκε με το θέμα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για το 2004 έχουμε ήδη τις πρώτες αποφάσεις και για, και για την οδηγία οδηγία του 2006 έχουμε ξεκινήσει την ε, ε, διαδικασία ε, Ελπίζουμε όμως να μπορέσουμε να τη διακόψουμε σύντομα γιατί τα κράτη-μέλη θα προβούν στα απαραίτητα μέτρα. Θα μιλήσω κυρίως για την οδηγία 2002 κάθετος 73 για την ισότητα της μεταχείρισης δηλαδή Υπήρξαν κάποιες διαδικασίες επί παραβάση που ξεκίνησαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 23 κράτη-μέλη για τα οποία ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, δρομολόγησε τη διαδικασία αυτή. Αυτή τη στιγμή παραμένουν 16 εκκρεμείς τέτοιου είδους διαδικασίες, κάτι το οποίο σημαίνει ότι καθ' όλη τη διάρκεια της περίοδου αυτής καταφέραμε μόνο 7 διαδικασίες επί παραβάση να ολοκληρώσουμε. Ε, θα σας μιλήσω για τις χώρες τις οποίες πρόκειται. Αυστρία, Φινλανδία, Κύπρος, Ελλάδα, Γαλλία, Μάλτα και Τσεχία. Σε αυτές τις επτά περιπτώσεις ε, λοιπόν ε, ολοκληρώθηκαν ε, οι διαδικασίες επί παραβάση κατόπιν τροποποίησης της νομοθεσίας που τελικά είχαν ως αποτέλεσμα να συνάδει νομοθεσία των κρατών μελών αυτών με την οδηγία και ε, μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις έχει ξεκινήσει η διαφαρμογή της οδηγίας. 16 ε, όμως διαδικασίες παραμένουν εκρεμείς και θα ήθελα να σας πω ότι στη μεγαλύτερη πλειοψηφία η τελευταία φάση της προκαταρτικής διαδικασίας έχει ολοκληρωθεί γιατί σε 14 περιπτώσεις ε, έχει έχουν ήδη αποσταλεί τα σχετικά στοιχεία και οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχουν σκοπό να περάσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας ε, Θα ληφθούν λοιπόν κατά τον επόμενο μήνα οι σχετικές αποφάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ή θα συνεχίσει η διαδικασία ε, επί παραβάση στο δικαστήριο ή θα κλείσει το θέμα αν συμμορφωθούν τα κράτη-μέλη, που αυτό ελπίζουμε να γίνει. Έχει, υπάρχουν όμως και πολλές άλλες οδηγίες, ε, εγώ επικεντρώθηκα σε αυτές τις τρεις. Ο υψηλός αριθμός ε, των διαδικασιών επί παραβάση σημαίνει ότι είναι ένα ζήτημα προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί όπως σας είπα, ο έλεγχος ε, της συμμόρφωσης και της ποιότητας της μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο είναι για μας μία προτεραιότητα. Όπως σας είπα και προηγουμένως, η προτεραιότητα αυτή ε, δίνεται στην πρώτη οδηγία 2002 κάθετος 73 ο έλεγχος της συμμόρφωσης ε, και της τη συμμόρφωση τη ε, οδηγία του 2002 και του 2004, ε, από ποιοτική απόψεως δηλαδή, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη, όμω θα ολοκληρωθεί στο δεύτερο εξάμεινο του 2010. Υπάρχει λοιπόν αυτή η ανάγκη να θέσουμε προτεραιότητες. Ο ένας λόγος είναι αυτός που σας ανέφερα προηγουμένως. Άλλος ένας λόγος είναι ότι αυτή η οδηγία του 2002 έχει, ε, συμπεριλαμβάνει πολλές αρχές ε, που ε, συμπεριλαμβάνονται και στις επόμενες οδηγίες του 2004 και του 2006. Επομένως, το να αξιολογήσουμε καλά την πρώτη οδηγία θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των διαδικασιών επί παραβάση που θα πρέπει να δρομολογήσουμε για τις μεταγενέστερες οδηγίες. Δεν ξέρω, ίσως να έδωσα πολλά αριθμητικά στοιχεία και πολλά... Σας ανέφερε ενδεχομένως πολλά γεγονότα. Και θα ήθελα ολοκληρώνοντας να πω ότι τα περισσότερα κράτη-μέλη έχουν επιτυχώς μεταφέρει την οδηγία. Θα ήθελα να συγχαρώ τα κράτη-μέλη για την προσπάθεια τους ε, αυτή. Όπως είπα, 16 διαδικασίες σε παραμένουν ανοιχτές ε, για την ισότητα της ε, μεταχείρισης και πρέπει να πούμε ότι ήταν δύσκολη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο. Και είναι προφανές, όπω είπε και η έκθεση, όπως ανέφερε και η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταφορά ε, της οδηγίας αυτής. Τα μέτρα που χρειάστηκαν ήταν αρκετά σημαντικά, γιατί κάποιες από τις διατάξεις είναι πάρα πολύ τεχνικές, το πεδίο εφαρμογής ε, ε, είναι αρκετά ευρύ και συνεπώς εξηγεί σίγουρα τα, τα αποτελέσματα αυτά. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο περιθώριο βελτίωσης και πρέπει να πω ότι τα κράτη-μέλη έχουν ακόμη πολλές προσπάθειες να καταβάλουν μέχρι να φτάσουν στην πλήρη συμμόρφωση με την οδηγία αυτή. Θα ήθελα επίση να πω ότι πάνω από το 1 τέταρτο των κρατών μελών ε, για τα οποία είχαν ξεκινήσει διαδικασίε επί παραβάση, εντωμεταξύ τροποποίησαν την ομοθεσία τους ε, με σκοπό τη συμμόρφωση. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ποτέ δεν ήταν βεβαίως ε, να διώξει ένα κράτος μέλος ε, ε, και να φτάσει στο δικαστήριο με τα κράτη-μέλη σε σχέση με την οδηγία αυτή και επειδή πολλά κράτη-μέλη ήδη συμμορφώθηκαν, ελπίζουμε ότι δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε ως εκεί γιατί και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη θα συμμορφωθούν. Ευχαριστώ πολύ. Στο όνομα της Επιτροπής μας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες αυτές. Είναι πολύ σημαντικό για μας να λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με το πώς εφαρμόζεται η που εκπονούμε εδώ. Είναι ένας τομέας που συχνά παραμελείται. Δείχνουμε μεγάλο ενδιαφέρον όταν έχουμε νέα θέματα και νέα νομοθεσία. Είναι πολύ σημαντικό όμως να ενημερωνόμαστε σχετικά με την παρακολούθηση της συνέχειας της νομοθεσίας. Είναι λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες σας. Ευχαριστούμε την Επιτροπή. Πρώτη ομιλήτρια, η κυρία Μπάουερ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που λάβαμε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για όσα άκουσα και για όσα δεν άκουσα. Όταν προκύπτει το ερώτημα αυτό, το θέμα της ισότητας των φύλων είναι πάντα το σημαντικότερο παράδειγμα. Δεν υπάρχει μόνο ένας σχετικός νόμος, υπάρχουν αρκετοί. Και επανειλημμένα αναφέρεται ότι οι νόμοι αυτοί θα πρέπει να εφαρμόζονται. Οι διατάξεις αυτές θα πρέπει να εφαρμόζονται. Αλλά αμφισβητείται πάντα η αποτελεσματικότητα από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι προφανώς επί Βελγικής Προεδρίας θα έχουμε μείωση των διαφορών, αλλά πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Πώς μπορούμε να πετύχουμε τέτοια εφαρμογή των διατάξεων, των νόμων, ώστε να μπορούμε να πούμε ότι είναι πραγματικά αποτελεσματική και ότι δεν υπάρχουν παραθυράκια. Η ερώτησή μου είναι, προβλέπονται αυστηρά μέτρα όσον αφορά τους νόμους αυτούς, διότι μου φαίνεται ότι θα πρέπει να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο. Χωρίς νέες νομοθετικές προτάσεις, μάλλον κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Δεν θα πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες. Δεν θα πρέπει να περιμένουμε ότι όλοι ξαφνικά θα γίνουν εργατικοί, θα αναλάβουν τις ευθύνες τους και ότι θα εφαρμοστούν πιστά όλοι οι νόμοι. Θα πρέπει να κάνουμε ένα βήμα προς τα μπροστά, ένα βήμα προόδου. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι δεσμευτικές οι διατάξεις, θα πρέπει να προβλέπονται κυρώσει σε περίπτωση που δεν πληρούνται. Θα μπορούσε να φανταστεί κανείς εισαγωγή τέτοιων μέτρων και θα ήθελα να ξέρω τι μπορούμε να περιμένουμε. Μία δεύτερη σημαντική ερώτηση κατά τη γνώμη μου. Το θέμα της ισότητας. Υπάρχουν διάφορες αρμοδιότητες που σχετίζονται με το θέμα αυτό σε πολλά κράτη-μέλη. Είναι αδιανόητο να πληρούνται απόλυτα αυτές οι διατάξεις, να εφαρμόζονται απόλυτα ισότητα και σε πολλές περιπτώσεις οι δυνατότητες για κάτι τέτοιο είναι πολύ περιορισμένες, ώστε να μην μπορούμε να μιλάμε για ισότητα στην πράξη. Υπάρχουν κάποια θετικά παραδείγματα. Σε πολλές περιπτώσεις έχουμε δει εφαρμογή, όχι όμως σε όλες. Δεν υπάρχει πάντα η δυνατότητα να γίνει κάτι τέτοιο και γι' αυτό θα ήθελα η Κομισιόν να μου πει τι μπορούμε να περιμένουμε στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Μπάουερ. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής έχει άλλες παρατηρήσεις. Δίνουμε το λόγο στον κύριο Περέιρα, παρακαλώ. Ορισμένα στοιχεία απάντησης προς την κυρία Μπάουερ. Όσο αφορά την, την ε, περίπτωση των αμοιβών, δεν ε, το ανέφερα, διότι όπως είπατε δεν είναι θέμα, δεν πρόκειται για θέμα μεταφοράς ή μετάταξης. Πρόκειται για το κατά πόσο οι κοινοτικοί κανόνες όπως ε, ισχύουν έχουν προσαρμοστεί έτσι ώστε να μην υπάρχει χάσμα αμοιβών. Εσείς πήρατε πρωτοβουλία για μια έκθεση σε αυτό το τομέα, γνωρίζετε πολύ καλά την κατάσταση, η ίδια η Κομισιόν πρότεινε στην ανακοίνωσή της ως προς το χάσμα των αμοιβών να σκεφτεί την αποδοτικότητα της νομοθεσίας για να καταπολεμήσουμε το χάσμα αμοιβών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προβεί σε έναν απολογισμό αυτού του εγχειρήματος στα πλαίσια της στρατηγικής ισότητα ανδρών γυναικών που θα εγκριθεί, αν γνωρίζω καλά, μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Άρα θα υπάρχουν στοιχεία πληροφόρησης σε σχέση με την εργασία που έγινε και την ειχνηλάτηση αποτελεσματικής αντιμετώπισης. Η κυρία Μπάουερ μας έδωσε ορισμένα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε σε πολλές πηγές πληροφοριών που διαθέτουμε. Ως προς την διαφάνεια μισθών και την ενίσχυση των κυρώσεων είναι μέτρα που θα πρέπει να μας απασχολήσουν. Και εδώ θα πρέπει να διαβουλευτούμε με τους κοινωνικούς εταίρους διότι η διαβούλευση με τους εταίρους είναι υποχρεωτική στα πλαίσια μιας τέτοιας πρωτοβουλίας. Ως προς τα equality bodies υπάρχει ένα πρόβλημα μεταφοράς οδηγίας σε ορισμένα κράτη-μέλη. Δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά ε, δυστυχώς ε, δεν, υπάρχει, ε, δεν υπάρχουν επαρκείς αρμοδιότητες από τα κράτη-μέλη ως προς τα equality bodies και θα ήθελα να πω ότι συμμερίζομαι την απόψή σας. Θα θέλαμε να δούμε ποιες είναι συγκεκριμένες αρμοδιότητες και θα πρέπει να γίνει μια διασαφήνιση για την αξιοπιστία και την αυτοδυναμία αυτών των οργανώσεων. Η Κομισιόν έχει ε, διενεργήσει μία μελέτη, διενεργεί μία μελέτη. Δεν έχουμε ακόμα τα αποτελέσματα για αυτούς τους φορείς, αλλά νομίζω ότι θα έχουμε μία καλύτερη θεώρηση της κατάστασης στα κράτη-μέλη, ιδιαίτερα ως προς τους ανθρώπινους σπόρους, αλλά και τους σπόρους γενικότερα για να δούμε πώς πρέπει να ανταποκριθούμε, ποιο είναι το επίπεδο επίβλεψης που προβλέπετε, γιατί πρόκειται για συλλογή δεδομένων. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το κείμενο της οδηγίας ε, σε σχέση με αυτούς τους φορείς δεν είναι τόσο σαφές. Και ίσως υπάρχει και θέμα μιας νομικής ανεπάρκειας. Μετά τη μελέτη θα δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε πώς μπορούμε, μετά την ε, μελέτη θα δούμε πώς θα ενισχύσουμε το ρόλο αυτών των οργανισμών ισότητας. Σας ευχαριστώ θερμά. Φτάσαμε Ολοκληρώσαμε τα θέματα που είχαμε στην ημερήσια διάταξη σήμερα. Θα διακόψουμε σύντομα και θα τα ξαναπούμε 5 και 4 για να συζητήσουμε την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Σύντομο διάλειμμα. Πριν διακόψουμε όμως θα ήθελα να θυμίσω στους συναδέλφους ότι αύριο είμαστε σε άλλη αίθουσα συνεδριάσεων. ΑΣΠ 3Ε2 παρακαλώ τους βουλευτές να μην αφήσουν εδώ τα έγγραφά τους μετά την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ στις 5 και 4. Σύντομο διάλειμμα μέχρι τις 5 και 4.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 Er- Στο όνομα της Επιτροπής μας, σας καλωσορίζω στην κοινή συνεδρίαση της Επιτροπής Ισότητας και της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Πολύ σημαντικό θέμα είναι η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Εισαγωγικά πολύ πολύ σύντομα να σας πω ότι 12 κράτη-μέλη έχουν παρουσιάσει πρωτοβουλία για μια οδηγία για την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας, η οποία παρουσιάστηκε στις αρχές της χρονιάς στο Συμβούλιο. Καθότι η προστασία θυμάτων, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για βία εις βάρος των γυναικών, καθώς και εις βάρος νέων κοριτσιών, που είναι σημαντικό κομμάτι του θέματος αυτού. Το θέμα αυτό εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και της Επιτροπής Ισότητας και γι' αυτό είναι πολύ καλό το ότι μπορούμε τώρα να συνεργαστούμε μεταξύ μας, να συνεργαστούν δηλαδή αυτές οι δύο επιτροπές που είναι αρμόδιες για το θέμα. Ισχύει ο κανόνας 51, ο που ρυθμίζει τη συνεργασία αυτή. Η σημερινή συνεδρίαση είναι η πρώτη κοινή συνεδρίαση για το θέμα αυτό. Και μοιράζομαι την Προεδρία με την κυρία Κιονέτ, που είναι η Πρόεδρος ε, της ε, Επιτροπής πολιτικών ελευθεριών και θα ήθελα να της δώσω τη δυνατότητα να εκφράσει τις θέσεις της πρωτού να δώσουμε το λόγο στην Ισπανική Προεδρία και στην Κομισιόν. Πρώτα λοιπόν να δώσω το λόγο στην κυρία Κίνγα Γκιόνς. Παρακαλώ. Um, thank you uh, Ευχαριστώ. Πριν αρχίσουμε τη συζήτηση επί της ουσίας του ζητήματος, θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και τη χαρά μου για το γεγονός ότι έχουμε αυτήν την κοινή συνεδρίαση, κάτι το οποίο συμβολίζει επίσης τη σημασία του θέματος αυτού, δεδομένου ότι είναι συνάδελφοι από την Επιτροπή Γυναικών και από την Επιτροπή Ελευθεριών του Πολίτη. Πρόκειται για ζητήματα που μας απασχολούν όλους. Η εντολή προστασίας αναφέρεται στα θύματα κάθε είδους βίας επί τη βάση του φίλου σε θύματα βίας επίσης, γενικότερα, και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε μια σφαιρική θεώρηση. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η σημερινή μας συνεδρίαση που είναι η κοινή. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά και δίνω το λόγο στην Ισπανική Προεδρία, τον κύριο Μολίνο Σκόβο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ για να σας παρουσιάσω αυτή την πρωτοβουλία που προκύπτει από την Ισπανική Προεδρία και άλλες 11 χώρες μέλη. Πρόκειται λοιπόν για μια πρωτοβουλία 12 κρατών μελών. Η βάση της πρότασης οδηγίας είναι η εξής. Τα μέτρα προστασίας σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν και αφορούν και αφορούν το 90, κατά το 90% των περιπτώσεων γυναίκες. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών δίνει τη δυνατότητα μιας σωστής εμπεριστατωμένης συζήτησης για το θέμα. Σήμερα υπάρχει μία διάκριση. Γιατί όλα αλλάζουν από τη στιγμή που ένα θύμα ενός αδικήματος περνάει τα σύνορα. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο σήμερα για την επέκταση της προστασίας του προσώπου αυτού πέρα από τα σύνορα του κράτους στο οποίο του χορηγήθηκε αυτή η προστασία. Και αυτό είναι κάτι το πραγματικά παράλογο. Πρέπει οπωσδήποτε να επιληθεί το ζήτημα αυτό, γιατί σήμερα κάθε πολίτης έχει πλήρη ελευθερία να μετακινείται από το ένα κράτος μέλος στο άλλο. Πιστεύουμε λοιπόν ότι τέτοιου είδους μέτρα πρέπει να εγκριθούν από τις εθνικές αρμόδιες αρχές. Συχνά πρόκειται για ποινικά μέτρα άλλες φορές για αστικά μέτρα, όμως ο στόχος είναι ίδιος. Να εξασφαλίσουμε ότι το θύμα δεν θα υποστεί ένα ακόμη αδίκημα. αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε κατά πόσο θα ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι το θύμα. Λαμβάνω υπόψη το γερμανικό σύστημα. Δηλαδή κάποιος που παραμένει στη Γερμανία, είναι Γερμανός ε, υπήκος και μεταβεί στην Ισπανία, δεν έχει σημασία κατά πόσο πρόκειται για ποινικό ή αστικό. Θα πρέπει να προστατεύεται στην Ισπανία. Μπορεί να περάσει διακοπές ε, ένα-δύο μήνες ή να έχει άδεια διαμονής, παραμονής έξι μηνών. Αυτό που έχει σημασία είναι το μέτρο να ισχύει και στην Ισπανία. Και αυτό ζητά το θύμα από τη Γερμανία. Διότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει σημασία εάν πρόκειται για αστικό ή ποινικό. Σημασία έχει η προστασία, η προστασία του φυσικού προσώπου. Δηλαδή να μην διαπραχθεί ένα νέο δίχημα και να μην υπάρχει αυτός ο βαθμός ευαλωτότητας επειδή το φυσικό αυτό πρόσωπο μετέβει από μία χώρα στην άλλη σε σχέση με το που διαπράχθηκε το δίκημα, Άρα βασιζόμαστε στο άρθρο 82 της νέας συνθήκης. Επίσης, πρόσφατα στο κείμενο υπάρχουν ορισμένες πιο διευρυμένες ερμηνείες, έτσι ώστε εάν δεν δεχτεί κανείς το θεσμευτικό χαρακτήρα της νομικής βάσης, θα, λάβει, θα ληφθεί υπόψη αυτή η συνεργασία και στον τομέα του ποινικού, δυνάμει του άρθρου 82. Επιμένω για το ότι καταφέραμε να ενσωματώσουμε στο παρόν κείμενο όλα τα μέτρα δυνάμει του ποινικού ή του αστικού, διότι θέλουμε να αποφύγουμε ένα αδίκημα και επειδή μιλάμε για αυτή την αποφυγή, μιλάμε για συνεργασία στον ποινικό τομέα. Αυτά δυνάμει των άρθρων 82 και 88. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία, διότι αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να συζητήσουμε αυτό το θέμα μαζί σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να έχουμε την δυνατότητα να γνωμοδετήσετε και εσείς και να βελτιώσετε το κείμενο. Είμαι ε, σίγουρος ότι θα βελτιωθεί το κείμενο αφού περάσει από το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε αυτή τη ε, δυνατότητα. Γι' αυτό θέλουμε συνεργασία στην Ισπανική, κατά την Ισπανική Προεδρία. Βεβαίως υπάρχουν και πολλά εμπόδια, πολλά ε, προσκόμματα. η Ισπανική Προεδρία και τα κράτη-μέλη που μας υποστηρίζουν δεν μπορούμε να, παρά να σας πούμε αυτό. Θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα διαλόγου μαζί σας. Καταλαβαίνουμε ότι ε, δεν θα ε, πρέπει να αντιταχθούμε σε αυτό το κοινό μέσον. Θα πρέπει λοιπόν να ε, να γίνει ένα πρώτο βήμα, να ληφθούν τα πρώτα μέτρα, που δεν θα είναι και τα τελευταία έπονται και άλλα. Θα πρέπει όμως να γίνει αυτό το πρώτο βήμα και για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μιλάμε για αμοιβαία αναγνώριση μέτρων υποστήριξης και προστασίας, κάτι το οποίο δεν ίσχυε μέχρι τούδε. Γι' αυτό θα θέλαμε με αυτή τη δυνατότητα να προωθήσουμε έναν διάλογο. Το νέο κείμενο, πιστεύουμε στο νέο κείμενο, στη δυναμική του, και όταν αναλύσετε αυτή την πρόταση, ε, αναλύστε το παρόν κείμενο, το οποίο θα οδηγήσει σε μία συμφωνία στο Συμβούλιο, διότι υπάρχει πολύ καλή διάρθρωση με τη νομική βάση. Αν έχετε οποιαδήποτε εμφιβολία. Εμείς ως Ισπανική Προεδρία θα επανέλθουμε, θα το συζητήσουμε ε, μαζί σας, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι να δούμε ποια είναι η νομική βάση η οποία ενισχύει αυτή τη συνεργασία ιδιαίτερα στον τομέα των ποινικών διώξεων. Τέλος, θα ήθελα να σας πω ότι πρόκειται για μία ε, πρόταση που ενέχει συγκεκριμένους μηχανισμούς έτσι ώστε ο δικαστής να μπορεί να συνδυάσει ε, αστικά με ποινικά μέτρα. Και κατά την εκτέλεση δεν ε, μιλάμε για τα ίδια μέτρα, υπάρχει αυτή η απόκληση. Αυτό που έχει λοιπόν σημασία είναι να ισχύσει ένας μηχανισμός όπου να εφαρμοστούν παρόμοια μέτρα στην χώρα εκτέλεσης έτσι ώστε να είναι, δυνατή αυτή, να είναι δυνατός αυτός ο συνδυασμός μέτρων. Δεν θα ήθελα να υπερβώ το χρόνο μου. Γι' αυτό θα σταματήσω εδώ. Βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις και επιμένω ότι θα θέλαμε να το συζητήσουμε από κοινού. Και εάν η τελική απόφαση του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου δεν αρέσει την Κομισιόν, θα πρέπει να γίνει προσφυγή στο 10. Αλλά, εν περιπτώσει, θα πρέπει να έχετε και εσείς τη δυνατότητα να αποφασίσετε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε την Ισπανική Προεδρία για τις πληροφορίες αυτές. Δίνουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Κομισιόν, τον κύριο Γιώναταν Φαουλ. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλό απόγευμα. Η Κομισιόν προφανώς στηρίζει τον στόχο πίσω από την πρόταση αυτή. Ποιο θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε άλλο. Υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα και υπάρχει ανάγκη για ευρωπαϊκή νομοθετική λύση. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το θέμα αυτό. Αλλά θα πρέπει να είναι σωστή η λύση, διότι εάν δεν είναι, θα χαθούμε σε χρόνια ε, νομικών αντιδικιών και οι άνθρωποι που θέλουμε να, προστατεύσουν, να προστατεύσουμε θα κατηγορούν όλους μας που δεν πετύχαμε να ρυθμίσουμε σωστά τις λεπτομέρειες. Και οι λεπτομέρειες εδώ είναι εξαιρετικά σημαντικές. Η συνθήκη κάνει μια σαφή διάκριση ανάμεσα στο ποινικό και στο αστικό δίκαιο. Είχαμε τεράστιες συζητήσεις σε όλες τις χώρες μας σχετικά με την επικύρωση της συνθήκης της Λισαβόνας και ένα από τα θέματα σε πολλές από τις χώρες μας ήταν ο ακριβής ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους διάφορους αυτούς τομείς δικαίου με αποτέλεσμα να ισχύουν πολύ διαφορετικοί κανόνες στο αστικό δίκαιο από τη μία μεριά και στο ποινικό δίκαιο από την άλλη. Έχουμε άλλα συστήματα ψηφοφοριών, άλλα κράτη-μέλη συμμετέχουν στην νομοθεσία, ε, ανάλογα με το αν βρισκόμαστε στον τομέα του αστικού δικαίου ή του ποινικού δικαίου. Θα πρέπει λοιπόν να ρυθμίσουμε σωστά το θέμα αυτό. Και σε αυτόν το πολύ σημαντικό τομέα του, της Ευρωπαϊκής Προστασία, Προστασίας οι εθνικές μας παραδόσεις είναι διαφορετικές. Ε, σε κάποιες από τις χώρες μας είναι θέμα ποινικού δικαίου, ενώ σε άλλες χώρες είναι θέμα αστικού δικαίου. και ε, πολύ συχνά η ίδια υπόθεση επιπτυχεί στο αστικό και στο ε, ποινικό δίκαιο. Ε, θα πρέπει λοιπόν οι τεχνικές λεπτομέρειες να είναι σωστές. Ξέρω ότι είναι σχεδόν τροπή να μιλάει κανείς για νομικές λεπτομέρειες, για νομική τεχνική όταν μιλάμε για ένα τόσο σημαντικό θέμα, αλλά μετράνε. Θα πρέπει να έχουμε σωστή ρυθμίση, διότι αλλιώς σε ένα-δύο χρόνια όλη η δουλειά μας θα καταρρεύσει, διότι δεν θα λειτουργεί η νομοθεσία, το δικαστήριο θα αρνηθεί να το ακολουθήσει και ο κόσμος θα ε, προσφεύγει στο δικαστήριο όχι σε ε, ε, περιπτώσεις πολύπλοκες αλλά σε περιπτώσεις που προκύπτουν λόγω των, τεχνικών, των νομικών τεχνικών τυχών. Έχουμε λοιπόν το θέμα της πρόληψης ε, στα πλαίσια του ποινικού δικαίου για το οποίο υπάρχει άλλο άρθρο της συνθήκης ε, και, ή, ε, και έχουμε και τον αντίστοιχο τομέα στο αστικό δίκαιο όπου ισχύει άλλη σειρά κανόνων. Η πρότασή μας λοιπόν είναι να προχωρήσουμε με βάση την πρόταση που έκαναν μια σειρά κρατών μελών και να περιοριστούμε στις, στο ποινικό δίκαιο και στις αρχές επόμενης χρονιάς να υποβάλουμε πρόταση για το υπόλοιπο του πεδίου εφαρμογής, ώστε ο ευρωπαϊκός νόμος, το σύνολό του, και σωστά βασισμένος σε κανόνες της συνθήκης, να μπορεί να ανταποκριθεί στα προβλήματα που προκύπτουν. Έτσι θα έχουμε μία σειρά, πλήρη σειρά μέσων ώστε τα, ε, ώστε τα δικαστήρια στα κράτη-μέλη να μπορούν να ε, εφαρμόζουν σωστά το νόμο χωρίς ε, φόβο αντιδικιών για θέματα ευρωπαϊκού δικαίου, συντάγματος κλπ. Δεν είναι δύσκολο να γίνει. Απλά θέλει κάποιο χρόνο, διότι εμείς, όχι τα κράτη-μέλη, θα πρέπει να κάνουμε μια σωστή μελέτη αντικτύπου πριν την προετοιμασία των νομοθετικών προτάσεων. Θα το κάνουμε αυτό. Ε, σχεδιάζουμε λοιπόν να υποβάλουμε σχετική πρόταση με, τον, με την κανονική διαδικασία και να την υποβάλουμε σε εσά και στο Συμβούλιο στι αρχέ του 2011, ώστε κατά τη διάρκεια τη επόμενη χρονιά να έχουμε την πλήρη σειρά νομοθετικών μέσων. Οτιδήποτε άλλο, κατά τη γνώμη μας, θα ήταν επικίνδυνο. Επικίνδυνο για την ίδια νομοθεσία που μπορεί να ανατραπεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά επικίνδυνο και για τους εμπλεκόμενους ανθρώπους, δίδοντάς τους μια ψευδή αίσθηση ασφαλείας ότι αντιμετωπίζουμε το πρόβλημά τους, ενώ δεν το κάνουμε σωστά σύμφωνα με τον νόμο διακυβεύοντα έτσι το όλο εγχείρημα και αυτό μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε δικαστήριο, σε οποιοδήποτε κράτο μέλο Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, ανα πάσα στιγμή, ε, αν υπάρξει νομική προσφυγή. Α το αποφύγουμε αυτό λοιπόν, α κάνουμε ε, σωστή δουλειά, ε, κάνοντα διάκριση από τη μία μεριά ανάμεσα στο ποινικό δίκαιο, ε, από τη μία για την ποινική διαδικασία και από την άλλη ε, με το αστικό δίκαιο και την πρόληψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την Κομισιόν για τι ε, πληροφορίε αυτέ και θα δώσω τώρα το λόγο στην εισηγήτρια μας από στις εισηγήτριές μας από την Επιτροπή Ισότητας και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Προτού να δώσω το λόγο στην κυρία Χιμένες, θα ήθελα να θυμίσω στους συναδέλφους ότι έχουμε διαρμηνία μέχρι τις 6.30 ώρα. Δίνω το λόγο στην κυρία Χιμένες. Παρακαλώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο του Συμβουλίου, την Κομισιόν και όλους όσους παρευρίσκεστε σήμερα στη συνεδρίαση και όπως είπε και η πρόεδρος της ΛΥΜΠΕ, ε, πρόκειται για ένα πολύ ενδιαφέρον κοινό πλαίσιο συζήτησης. Βεβαίως αυτό μας ενδιαφέρει είναι η υπεράσπιση του θύματος. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι ο κόσμος του θύματος, ιδιαίτερα όταν μιλάμε για την ΕΤΑ και για τις τρομοκρατικές δραστηριότητες που οδηγούν σε σωρία θυμάτων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ζήσαμε ε, μεγάλες απώλειες στις ε, οικογένειές μας και εγώ προσωπικά. Γι' αυτό το Δεκέμβριο πέρσι στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης ε, παρουσίασα μία τροπολογία έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα, δηλαδή να απομακρύνουμε τον θήτη από το θύμα. Γι' αυτό ε, θέλησα να είμαι εισηγήτρια, κάτι το οποίο μου επετράπει το Μάρτιο και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε σε αυτή την εντολή προστασίας και ώστε να είναι αποτελεσματική. Έτσι ώστε όταν κάποιος προστατεύεται στη χώρα του, αυτόματα να μπορεί να προστατευτεί σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να επιληθεί αυτό το ζήτημα, αλλά δεν είμαι τόσο πεπισμένη γι' αυτό. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι η πρόταση προωθήθηκε από το Συμβούλιο, αλλά η Κομισιόν έθεσε τροχοπέδι, θεωρώντας ότι αυτό θέμα, το θέμα είναι δικής της αρμοδιότητας, η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας δηλαδή. Γι' αυτό έχουμε να κάνουμε με μια διχογνωμία μεταξύ Κομισιόν και Συμβουλίου. Το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να είναι όμοιρος όμως ούτε της Επιτροπής ούτε του Συμβουλίου. Δεν πρόκειται για οδηγία κανενός, ούτε η δική μου, ούτε της κυρίας Ρομέρο, ούτε της Κομισιόν. Πρόκειται για μια οδηγία που θα πρέπει να υπηρετεί τα θύματα. Θα πρέπει να βοηθήσει όλους τους ανθρώπους που θέλουν να μετακινηθούν ελεύθερα στην Ευρώπη για να έχουν το ίδιο επίπεδο προστασίας που έχουν στη χώρα τους. Θα πρέπει να εξεύρουμε μία λύση διότι αρμόζει στα θύματα. Εμείς υποστηρίζουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας. Δεν θέλουμε βεβαίως να δώσουμε μετάλλιο σε κανέναν θα πρέπει να φτάσουμε σε μια οδηγία που πραγματικά να προστατεύει το θύμα, τα θύματα. Να μην αφήσουμε τα θύματα χωρίς πραγματική προστασία. Χρειάζεται ουσιαστική προστασία για την καταπολέμηση της ανισότητας των δύο φύλων. Θα πρέπει να ισχύει σε όλες τις χώρες. Και θα ήθελα το Συμβούλιο να μου πει τι θα γίνει με το 9C που μιλά για χώρα εκτέλασης η οποία μπορεί να μην αναγνωρίσει το δίκημα από το οποίο διαπράχθηκε στη χώρα η οποία εξέδωσε την εντολή προστασίας. Αυτό που έχει σημασία είναι να προστατεύσουμε το θύμα τάχιστα με πλήρη αναγνώριση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα μέσο το οποίο να προστατεύει τα θύματα πλήρως, χωρίς να μπούμε σε μια πολεμική μεταξύ κρατών μελών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τη θέση του θύματος που έχει υποστεί κόποση. Δεν έχει πάντα τη διάθεση να δώσει μάχες. Γι' αυτό θα πρέπει να ε, βρούμε μία συνένεση, να προστατεύσουμε τα δικαιώματα του θύματος και να μην υπάρχουν εξαιρέσεις. Θα πρέπει να εγγυηθούμε αυτή την προστασία, γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστούν τα τρία ε, θεσμικά όργανα, διότι δεν έχει σημασία να απονείμουμε ένα μετάλλιο εδώ θα πρέπει να είμαστε ικανοποιημένοι διότι με βάση τη δική μας εργασία τα θύματα μπορούν να κινηθούν πολύ πιο ελεύθερα στην Ευρώπη. Γι' αυτό θα συνεχίσω να εργάζομαι για τα δικαιώματα των θυμάτων. Θα πρέπει αύριο να έχουμε μία εντολή που να είναι πιο φιλόδοξη, όπου να περιλαμβάνονται όλα τα θύματα, οι ανήλικοι, τα, του, τα θύματα της τρομοκρατίας, της μαφίας, της δουλεμπορίας και ούτω καθεξής. Θα πρέπει να μιλάμε ανοιχτά για θύματα και να βάλουμε το θύμα στην θέση που πραγματικά του αξίζει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Χιμένες θα ακούσουμε ε, τώρα την ε, αρμόδια η συγγήτρια από την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Παρακαλώ κυρία Ρομέρο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ζούμε μία πολύ σημαντική στιγμή γιατί για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποβάλλεται μία εντολή προστασίας για τις γυναίκες που πλήττονται και αποτελούν θύμα βίας. Ε, η εικόνα είναι ενθαρρυντική, διότι για πρώτη φορά μιλάμε για μία πραγματική βία κατά αυτών των γυναικών και για πρώτη φορά υπάρχουν δύο κράτη-μέλη που προέβαλαν αυτή την πρωτοβουλία. Αυτή η βία είναι παρούσα και στην εργασία μας, στην κοινοβουλευτική μας εργασία. Γι' αυτό πιστεύω ότι η πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου ήταν άκρος ενδιαφέρουσα, άκρος ευπρόσδεκτη από, τις όλες τις, από όλες τις οργανώσεις γυναικών και όλους όσους ανησυχούν για την κατάσταση των γυναικών. Και θεωρούμε ότι η Κομισιόν δεν έλαβε την πρωτοβουλία όπως και όποτε θα έπρεπε. Γιατί η Επιτροπή δεν είχε αναλάβει τα καθήκοντά της εκείνη τη χρονική στιγμή και γι' αυτό το Συμβούλιο υπέβαλε ένα πραγματικό πρόβλημα το, που, το οποίο ζούμε στις ευρωπαϊκές χώρες και γι' αυτό θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για μια κατάσταση κατεπήγοντος, για μια επίγουσα ανάγκη. Η Κομισιόν δεν είχε αναλάβει καθήκοντα τότε και έπρεπε την ε, πρωτοβουλία να προωθήσει το Συμβούλιο. Μιλάμε για μια πρόταση οδηγίας για τα θύματα της τρομοκρατίας αρχικά. Εδώ μιλάμε για θύματα όπου υπάρχει ένας θήτης ο οποίος έχει οριστεί, είναι γνωστός. Άρα το πεδίο εφαρμογής είναι πιο περιορισμένο από την αρχική οδηγία. και δεν αποτελεί τροχοπέδι για την οδηγία της Επιτροπής σε σχέση με τα θύματα τρομοκρατίας. Θεωρούμε ότι αυτή η οδηγία είναι ένα πρώτο βήμα και θα ήταν άκρος ενδιαφέρον να υπάρξει ποινική συνεργασία στον τομέα της πρόληψης. Είναι πολύ θετική η εικόνα, γιατί κάνουμε τα πρώτα βήματα για μία πρόληψη στο θέμα της ποινική συνεργασίας. Μιλάμε για γεγονότα που πολύ χαρακτηρίζουν ε, ίσονο σημασία, γιατί μιλάμε για βία που άπτεται των δύο ε, φύλων. Υπάρχουν πολλά τέτοια συμβάντα. Μιλάμε για κακομεταχείριση των γυναικών με ψυχικές επιπτώσεις που μπορούν να οδηγήσουν και στο θάνατο. Υπάρχει ο, μηχός, ο μηχανισμός καταγγελίας των γυναικών, αλλά πολλές φορές αυτά τα συμβάντα έχουν οδηγήσει και σε θάνατο. Θα πρέπει λοιπόν να αποτρέψουμε τους θανάτους. Γιατί το άρθρο 1 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μιλάει για ανθρώπινη και φυσική ακαιρεότητα. Δεν μιλάμε για θέματα ίσονος σημασίας, για μικροελήψεις ή κακή συνεννόηση μέσα στο ζευγάρι. Είτε πρόκειται για συζύγους είτε όχι. Ε, πρόκειται για ένα θέμα το οποίο ε, δυστυχώς δεν ε, συζητιόταν ανοιχτά σε πολλές χώρες. Γι' αυτό ζητήσαμε από ένα παρατηρητήριο να διενεργήσει μελέτες για να δούμε τι συμβάντα υπάρχουν και κατά πόσο μπορούν να αναγνωριστούν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τις εθνικές εντολές προστασίας και μπορούμε να κάνουμε μια προβολή, μια προεκβολή και μπορούμε να μιλήσουμε για εκατοντάδες χιλιάδες εντολές προστασίας. Μόνο στην Ισπανία έχουμε 102.000 τέτοιες εντολές όπου έχουμε 4.000 γυναίκες οι οποίες προέρχονται από την Ρουμανία και αποτελούν, έχουν αποτελέσει θύματα ή είναι ενδυνάμει θύματα. Υπάρχουν και περιπτώσεις ε, φόνων καθημερινά στην Ισπανία. Θα θέλαμε η Κομισιόν να γνωρίζει ότι μιλάμε για μια κατάσταση κατεπήγοντος, για μια επίγουσα ανάγκη. Το παρατηρητήριο του WAVE, Women Against Violence in Europe, μιλά για 2.500 θύματα στην Ευρώπη. Εάν λάβουμε υπόψη την εμβέλεια του προβλήματος και αν ορίσουμε ορισμένες παραμέτρους σε σχέση με τα θύματα τρομοκρατίας, θα μπορούσαμε να έχουμε παρόμοια αριθμητικά στοιχεία με αυτά που γνώρισαν η ΙΠΑ ε, το Σεπτέμβριο στις 11 Σεπτεμβρίου του 2009. Μιλάμε για ε, εφάμιλο αριθμό θυμάτων. Όλα αυτά έχουν κοινοβουλευτικό αντίκτυπο. Γι' αυτό ζούμε μία στιγμή ελπίδας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναλύσει το θέμα όπως αρμόζει, ίσως με μία διαφορετική οπτική γωνία, γιατί άλλα είναι τα θύματα ε, τρομοκρατίας ή θύματα γενικότερης ή άλλης βίας. Θα πρέπει όμως να διανοίξουμε το δρόμο για μια άλλη οδηγία που έχει κατά νου η Κομισιόν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως θα παρακολουθήσει αυτή την πρωτοβουλία λαμβάνοντας υπόψη τον διτό αυτό χαρακτήρα και θα ήθελα εν κατακλείδη να τονίσω μετά τις παρεμβάσεις της Κομισιόν και του Συμβουλίου ότι ως προς αυτό το θέμα θα ήταν ε, λυπηρό να σφάλουμε. Γιατί μπορούμε να αποφύγουμε την ύπαρξη ορισμένων θυμάτων. Ίσως το δικαστήριο του Λουξεμβούργου δώσει άλλη ερμηνεία, αλλά εάν η Ευρωπαϊκή Εντολή Προστασίας τεθεί σε εφαρμογή, θα μπορέσουμε να αποφύγουμε μελλοντικά θύματα. Γι' αυτό θα πρέπει <coughs> να τηρήσουμε τις προθεσμίες, να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση που ανέκυψε με μέτρα που είναι περίπλοκα, που θα πρέπει να αναλυθούν λεπτομεριακώς, αλλά νομίζω ότι με τη συνεργασία του Κοινοβουλίου θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα που όρισε, τα προβλήματα που όρισε και η άλλη εισηγήτρια και με την κοινοβουλευτική μας εργασία θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το κείμενο και θα βελτιώσουμε και περιθωριακά ζητήματα που άπτονται του κεντρικού. Ευχαριστώ κυρία Ρομέρο. Τρεις συνάδελφοι ζήτησαν το λόγο. Εάν υπάρχουν άλλοι που έχουν απόψεις, και θέλουν να συμμετάσχουν στη συζήτηση, καλό θα είναι να ζητήσετε το λόγο. Οι τρεις που τώρα βρίσκονται στον κατάλογο των ομιλητών είναι ο κ. Μπούσετιλ, η κυρία Μπόσκοιτ και η κυρία Μπιλμπάου. Ε, οι υπόλοιποι που θα ζητήσουν το λόγο θα ε, εγγραφούν στον κατάλογο των ομιλητών. Να σας θυμίσω ότι έχουμε περιορισμένο χρόνο στη διάθεσή μας. Δίνω το λόγο πρώτα στον κύριο Πουστήλ. Yes, thank you, Madam. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστώ και τους δύο μιλητές ε, για την παρουσίασή τους. Εγώ είμαι συντονιστής εκ μέρους ε, της ομάδας του ΕΛΚ ε, και εκ μέρους Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και θα ήθελα να πω ότι είμαι κάπως απογοητευμένος από αυτά που παρουσιάζονται και ειδικότερα την ε, διοργανική πτυχή του θέματος αυτού μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Είναι, με μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Συμβούλιο μας λέει πάρετε την πρότασή μας ε, και εγκρίνετε την ε, το συντομότερο δυνατόν. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει «Α, ε, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένη με την πρόταση αυτή, εμείς δεν είμαστε ευχαριστημένοι με την πρόταση αυτή και πρέπει να πάμε στο δικαστήριο για να την αλλάξουμε». Κάνετε δηλαδή ό,τι μπορείτε, φλερτάρετε μαζί μας ε, και οι δύο πλευρές για να μπορέσουμε να εγκρίνουμε την πρόταση. Κοιτάξτε, δεν βρίσκω ότι είναι σοβαρά πράγματα αυτά και συγγνώμη που λέω προς τον ομιλητή από το Συμβούλιο, να το κάνουμε αυτό και μετά να τους αφήσουμε να μας πάνε στο δικαστήριο. Ε, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Και το ίδιο έχω να πω και προς τον κύριο Φολ. Γιατί το να εγκρίνουμε μία προσέγγιση που τα περιορίζει όλα μόνο στο ποινικό κομμάτι, όπως είπατε κι εσείς, ουσιαστικά σημαίνει ότι η νομοθεσία αυτή θα ισχύει μόνο για μερικά κρατημέλη. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να προχωρήσουμε. Εγώ θα έλεγα ότι και τα δύο όργανα θα έπρεπε να ξαναρχίσουν από την αρχή και να βάλουν τάξη στην πρότασή τους, να συμβιβαστούν, να συμφωνήσουν και να επανέλθουν ενώπιόν μας με κάτι το οποίο παρουσιάζει μία συνοχή, γιατί για την ώρα δεν ισχύει αυτό. Είναι θλιβερό, θλιβερότατο, είναι η δεύτερη φορά που βρισκόμαστε ενώπιον αυτής της κατάστασης, ε, δηλαδή διαφωνία μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Διερμηνία και μετάφραση ήταν το άλλο θέμα. Ακόμη και εκεί μπορούσαμε να νιώσουμε την ένταση μεταξύ του Συμβουλίου που είχε τη δική της πρόταση και μετά και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που στη συνέχεια ακολούθησε με την δική της ξεχωριστή πρόταση σωστό είναι αυτό όταν χρησιμοποιούμε αυτήν την ε, νέα εξουσία που μας δίνει η συνθήκη και που δίνει τη δυνατότητα και στο Συμβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχουν το δικαίωμα της πρωτοβουλίας. Δεν νομίζω ότι είναι ο σωστός τρόπος χρήσης αυτού του δικαιώματος πρωτοβουλίας και δεν νομίζω ότι μας βοηθάει ιδιαίτερα σε σχέση με αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Προτείνω λοιπόν να ζητήσουμε νομικές συμβουλές από τη νομική υπηρεσία μας για να μας καθοδηγήσει κάποιος και να μας πει ποια ακριβώς είναι η κατάσταση από νομική απόψεως. Πρέπει να ακολουθήσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο. Ποιος έχει δίκιο, εν πάση περιπτώσει. Οπωσδήποτε λοιπόν θα ζητήσουμε Συμβουλέ και καθοδήγηση από την νομική υπηρεσία και στη συνέχεια θα καταλήξουμε σε κοινή απόφαση, γιατί εδώ είναι συναρμόδιες δύο επιτροπές, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να βιαστούμε, να εγκρίνουμε μία νομοθεσία όταν υπάρχει σαφής απειλή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, «Ω, θα σας πάω στο δικαστήριο». Επ' αυτού δεν νομίζω ότι είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Μπόσκουρτ. Ευχαριστώ πολύ. Κοιτάξτε, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι μια πολύ καλή πρόταση. Θα έπρεπε να υπάρχει μια ευρωπαϊκή εντολή προστασίας, αλλά νομίζω επίσης ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί μήπως δεν μπορεί τελικά να εφαρμοστεί λόγω κάποιων ε, προβλημάτων. Πρέπει να κάνουμε λοιπόν καλά τη δουλειά μας. Αυτό είναι το χρέος μας προς τις γυναίκες που απειλούνται. Κοιτάξτε, μπερδεύτηκα λιγάκι. Όταν η πρόταση παρουσιάστηκε, αναφέρθηκε ότι σκοπό είχε να προστατεύσει τις γυναίκες. Μετά ακούσαμε ότι ήταν για όλους. Και τώρα επανερχόμαστε στο επιχείρημα ότι είναι πάλι για τις γυναίκες. Δεν καταλαβαίνω τελικά, αφορά συγκεκριμένα τις γυναίκες ή όχι. Και έχω ένα ακόμη ερώτημα. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας λέει ότι ισχύει μόνο για ε, ποινικά αδικήματα. Τι ακριβώς εννοείται. Θα ήθελα να μου το καταστήσετε λίγο πιο συγκεκριμένο. Η παρενόχληση ας πούμε. Και εφόσον είπατε ότι είναι πρόταση των 12 κρατών μελών, υπάρχουν 15 άλλες που δεν συμμετείχαν τόσο στην παρουσίαση αυτής της πρωτοβουλίας. Δηλαδή, οι υπόλοιπε 15 χώρε δεν συμφωνούν. Θέλαμε να μα πείτε λίγο περισσότερα για την ισορροπία δυνάμεων στο Συμβούλιο και θα ήθελα επίση να εκφράσω την ελπίδα μου ότι θα τα καταφέρετε και ότι θα παρουσιάσετε μια καλή πρόταση για να μπορέσουμε κι εμεί να βοηθήσουμε πραγματικά τι γυναίκε που χρειάζονται απεγνωσμένα την βοήθεια αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καταρχήν, θα πρέπει να σας πω ότι η βραχία μου ε, πήρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, σχετίζεται με θέματα τα οποία με, θέματα που με απογοήτευσαν, διότι μια τέτοια πρωτοβουλία θα, δεν θα έπρεπε να ε, οδηγείται μάλλον να αποτελεί απότοκο μίας ε, κατάστασης διχογνωμίας. Δηλαδή, με ποιος θα συνταχθούμε, με, το, με την Κομισιόν ή με το Συμβούλιο. Φαίνεται ότι δεν στοιχίζει τίποτα να φωνεύονται γυναίκες στην Ευρώπη. Γιατί αυτή είναι η πεμπτουσία του διλήμματος. Αλλιώς θα είχαμε φτάσει σε μία απόφαση. Πιστεύω ότι είναι μία πολύ καλή πρωτοβουλία. Νομίζω ότι θα πρέπει να βρούμε μία λύση έτσι ώστε οι γυναίκες και οι άνδρες να τύχουν προστασίες διότι στον 21ο αιώνα και με τη νομοθεσία που έχουν τα διάφορα κράτη-μέλη θα έπρεπε να ενταχθεί και μία νέα πραγματικότητα. Δηλαδή να λάβουμε υπόψη και τους ε, ομοφιλοφίλους που πλήττονται από τέτοιες μορφές βίας. Θα έπρεπε λοιπόν να συμπεριλάβουμε και αυτή την πραγματικότητα. Επειδή η εικόνα δεν είναι επιθυμητή, θα πρέπει να εγκρίνουμε κάτι το απτό για να βοηθήσουμε τις γυναίκες θύματα αλλά θα ήθελα να διατυπώσω μία ερώτηση προς το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Βλέπετε, διαβλέπετε κάποια δυνατότητα εξέβρεσης λύσης και αυτό είναι περισσότερο μία έκκληση. Μπορούμε να φτάσουμε σε μία λύση μέσα στη προθεσμία, στα πλαίσια της προθεσμίας που διαθέτουμε, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τις γυναίκες και τους άνδρες να μπορούν να τύχουν προστασίας από την ε, οικιακή βία βραχυπρόθεσμα ή αν δεν είναι δυνατόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταβάλει μια προσπάθεια έτσι ώστε να ενσωματώσει αυτή την προσωρινή λύση στην πρότασή της για το 2010. Διαφορετικά, όχι μόνο δεν προστατεύουμε τις γυναίκες, αλλά δημιουργούμε μεγάλη ανασφάλεια στις γυναίκες γιατί οι γυναίκες δεν μπορούν να προσφύγουν σε αυτή την εντολή. Άρα δεν έχουμε συνεισφέρει στην προστασία αυτών των ευάλωτων ανθρώπων. Ευχαριστώ. Να σας θυμίσω ότι πολλές ερωτήσεις τίθενται προς την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Η θα παρακαλούσα λοιπόν τους τέσσερις ομιλητές που έχουμε στον κατάλογο να είσαστε σύντομοι, ώστε να προλάβουμε να ακούσουμε την απάντηση της Κομισιόν και του Συμβουλίου. Κύριε Κώστα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι ένα θέμα ύψης της σημασίας. Είχαμε 12 κράτη-μέλη και μετά μία πλειοψηφία στο Συμβούλιο που θέλησε με αυτή την ε, πρωτοβουλία να καλύψει ένα νομικό κενό το οποίο είχαμε αισθανθεί ιδιαίτερα. Όχι μόνο εμείς οι γυναίκες, οι Ευρωπαίες γυναίκες, αλλά και θύματα, οι ενδυνάμει θύματα που δέχτηκαν σοβαρές απειλές. Αυτό αφορά και τους ε, ανηλίκους θα πρέπει να εποπτεύσουμε και την κατάσταση των ανηλίκων. Δέχομαι και συμμερίζομαι αυτά που είπε η συνάδελφος Ρομέρο, διότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να προσδώσει την δέουσα ε, προσοχή σε αυτό το θέμα, έτσι ώστε να μην υπάρχει διχογνωμία και ε, ρήξη αρμοδιοτήτων μεταξύ Συμβουλίου και Επιτροπής. Πρόκειται για έναν ε, επιθυμητό στόχο και έχουμε καθήκον ως βουλευτές να προωθήσουμε αυτή τη δράση τηρίζοντας και, τηρώντας, με συγχωρείτε, και υποστηρίζοντας και τις καινοτομίες που απορρέουν από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Διότι αυτό που έχει σημασία είναι η ελεύθερη κυκλοφορία προσώπων, η ασφάλεια των φυσικών προσώπων, η προστασία των γυναικών, η καταπολέμηση της δουλεμπορίας των γυναικών, όλα αυτά θα πρέπει να τύχουν της προστασίας μας κατά τον πλέον διεξοδικό τρόπο. Δεν θα πρέπει το άρθρο 82 να τύχει μιας συσταλτικής ερμηνείας. διότι οι δικαστικές αρχές θα μας συνδράμουν σε αυτή την εντολή προστασίας. Όπως είπε και το Συμβούλιο, θα πρέπει να δούμε κατά πόσο δεν υπάρχει η δυνατότητα να ερμηνεύσουμε αυτό το άρθρο λιγότερο συσταλτικά έτσι ώστε οι αρμόδιες αρχές ε, να μπορέσουν να το αντιμετωπίσουν καταλληλότερα τους συνδέοντα. Δεν μιλάμε για εναρμόνιση του, του δικαστικού τομέα. Απλώς οι δικαστικές αποφάσεις θα πρέπει να εφαρμόζονται παντού. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα διοικητικά δικαστήρια, τα αστικά και τα ποινικά. Αλλά οι αποφάσεις είναι δικαστικές αποφάσεις που θα πρέπει να τηρούνται παντού, έτσι ώστε να μην υπάρχει ανισορροπία προστασίας. Αυτή είναι μια έκκληση προς την Επιτροπή. Θα πρέπει υπό το φως της συνθήκης της Λισαβόνας να προχωρήσουμε προς τα εμπρός μέσα στα πλαίσια της ατζέντα μας, της κοινής ατζέντα των Επιτροπών ΛΥΜΠΕ και ΦΑΜ. Και θα θέλαμε να ζητήσουμε και την ε, γνώμη της Νομικής Επιτροπής του Κοινοβουλίου. Θα πρέπει οι συντονιστές να ασχοληθούν με αυτό το ζήτημα, όπως ζήτησε και το ΕΛΚ. Θα πρέπει να υπάρχει η μέγιστη δυνατή προστασία προς τις γυναίκες, προς τα θύματα. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όχι η συσταλτική ερμηνεία του δικαίου. Ας δούμε το περιεχόμενο των αγαθών που θέλουμε να προστατεύσουμε. Ευχαριστώ. Η κυρία Μοβάη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στη νομική σχολή είχα καθηγητή που έλεγε ότι δικηγόρος γίνεσαι όταν βρίσκεις τη σωστή λύση σε νομικό δίλημα και όταν βρεις ποια είναι η σωστή λύση, να βρεις τη νομική λύση που να στηρίζει αυτό. Η ερώτηση λοιπόν είναι, θέλουμε να προστατεύσουμε αυτές τις γυναίκες και αυτούς τους άντρες. Και αν ναι, και ελπίζω πραγματικά η απάντηση να είναι ναι, διότι είμαι δικηγόρος ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα τα τελευταία 25 χρόνια και έχω να κάνω με ε, ε, θύματα. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι να βρούμε τη σωστή λύση. Θα πρέπει να απελευθερώσουμε το θέμα αυτό από το κλουβί του να το βλέπουμε σαν ε, ένα θέμα ε, τεχνικής ε, συνεργασίας στον τομέα του ποινικού δικαίου. Δεν είναι. Και δεν είμαι φανατική θαυμάστρια της συνθήκης της Λισαβόνας, αλλά μια και την έχουμε, ας χρησιμοποιήσουμε την ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα δημιουργικά προς όφελος των επιζώντων και των θυμάτων. Και μια... Έχω και μια τεχνική ερώτηση. Μια ένα από τα συμπεράσματα της πρότασης είναι ότι τα θύματα ή οι επιζώντες ή τα πιθανά θύματα θα πρέπει να λαμβάνουν το ίδιο είδος προστασίας στο εξωτερικό όπως και στη δική τους χώρα. Πώς είναι δυνατόν τεχνικά σε περιπτώσεις όπου για παράδειγμα η κυρία Σβένσον, η ε, πρόεδρος της Επιτροπής Γυναικών ε, έχει, έχει συμπεριφερθεί ε, επαναστατικά έχει αναφέρει τις δικές της εμπειρίες. Στη Σουηδία έχετε σύστημα με ηλεκτρονικό βραχιόλι, αλλά στην Ουγγαρία όσοι επιβιώνουν, επιζούν σε περίπτωση οικιακής βίας, τι θα κάνουμε, τι, θα κάνουμε όσον αφορά την τεχνολογία και στο τέλος συνεδρίασης θα ήθελα να δώσω την αθοδέσμη αυτή στην κυρία Σβένσον ε, εκ μέρους ε, των γυναικών ε, που βοηθήθηκαν από το ότι τους εξιστορήσατε στην μέρα των γυναικών την πολύ θλιβερή ιστορία σας αλλά και την ιστορία των επιτυχιών σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ στο τέλος της συνεδρίασης. Θα σας δώσω την αθοδέσμη. Ehm, σας ευχαριστώ θερμά. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιανακουδάκη είναι η επόμενη ομιλήτρια. Παρακαλώ. Um, ευχαριστώ. Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι υπάρχει ανάγκη για το μέσο αυτό και υπάρχει και μια βασική ανάγκη, όπως είπε το Συμβούλιο. Συμφωνώ με την έκκληση να κάνουμε εμεί τα πρώτα βήματα. Αυτό θα ήταν πολύ ωραίο, ε, εφόσον είναι εφικτό. Η βία δεν έχει σύνορα, το ξέρουμε αυτό. Θέλουμε να στηρίξουμε την πρόταση αυτή, ωστόσο, ανησυχώ ότι υπάρχει διάσταση απόψεων σχετικά με το πού βρισκόμαστε από νομικής πλευράς. Πιστεύω ότι μπορούμε να ε, πάρουμε τα πρώτα να κάνουμε τα πρώτα βήματα, αλλά θα αποτύχουμε αν δεν ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα τώρα. Πολλού τομεί δεν έχουμε καλύψει. Θα πρέπει νομικά να βρούμε που στεκόμαστε. Ε, μιλάμε για ποινικό δίκαιο. Τι θα, τι θα κάνουμε με το αστικό δίκαιο, διότι... Πράγματι, ε, η πρόταση αυτή θα ισχύει μόνο σε κάποια κράτη-μέλη και όχι σε άλλα. Οι γυναίκε, λοιπόν, θα έχουν μια ψευδή αίσθηση ασφαλείας, ε, θα κάνουμε περισσότερη ζημιά αν υιοθετήσουμε την πρόταση αυτή στο παρόν στάδιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί βιαζόμαστε εφόσον υπάρχουν όλοι αυτοί οι τομείς που βρίσκονται ακόμα υπό συζήτηση. Θα ήθελα περισσότερο χρόνο. Σα ζητώ λοιπόν γιατί βιαζόμαστε. Θα υπάρχει το πρόβλημα και αύριο. Αν όμως το αντιμετωπίσουμε σωστά, θα το αντιμετωπίσουμε μια και καλή. δεν θα αλλάζουν χώρα οι γυναίκε και θα πιστεύουν ότι προστατεύονται, ενώ δεν προστατεύονται στην πραγματικότητα επειδή πρόκειται για ποινικό θέμα και όχι αστικό. Ε, θα πρέπει να ξέρουμε ποιο είναι το πεδίο εφαρμογή. Ε, η πρόταση θα καλύπτει τι γυναίκε, θα καλύπτει όλου. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι ευρύ το πεδίο εφαρμογή, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε ε, τα παιδιά και του άντρε ακόμα. Θα ήθελα η Κομισιόν και το Συμβούλιο να συμφωνήσουμε. Δεν έχει νόημα να απειλεί ο ένας τον άλλον με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό είναι πεδαριώδες. Βρείτε τα παραθυράκια, βρείτε τις αδυναμίες της πρότασης ε, και ας ε, δημιουργήσουμε ισχυρή νομοθεσία η οποία θα πετύχει το στόχο της. Μέχρι τότε όμως σας περιμένουμε. Το λόγο έχει η κυρία Γκόμες. Παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ υποστηρίζω την ανάγκη του να προχωρήσει αυτή η πρόταση. Και δεν καταλαβαίνω ακριβώ ποιο είναι το πρόβλημα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν έχει συγκεκριμένε αντιρρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγώ θα ήθελα να μα τι πει. Γιατί η διάκριση μεταξύ αστικής και ποινική ε, διαδικασίας δεν μου φαίνεται επαρκής ε, για να συνεχίζει ή να, να μην συνεχίζει εν πάση περιπτώσει η, η, η πρόταση αυτή. Άκουσα και την άποψη τη Βρετανική. Το γεγονός ότι οι εντολές προέρχονται από το αστικό δίκαιο δεν σημαίνει ότι αν είναι ποινικό το αδίκημα στο πλαίσιο αυτή της εντολής δεν μπορεί να προχωρήσει. Πρέπει να δούμε πώς ακριβώς λειτουργεί. Δηλαδή το ένα δεν προκύπτει από το άλλο. να δούμε, εν πάση περιπτώσει, πώ μπορεί να συμμορφωθεί όλο αυτό με τα διάφορα νομικά μα ε, συστήματα. Πέρα από αυτό όμω, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το Συμβούλιο, γιατί υπάρχει κάποια σύγχυση. Κάποια κράτη-μέρη ασχολούνται με αυτό το ζήτημα της, ε, των γυναικών ε, ως θυμάτων βίας κλπ. κλπ. Δεν αφορά όμω μόνο τις γυναίκες, αφορά όλους όσους έχουν ανάγκη και ε, ήταν αντικείμενο... Ε, ήταν θύμα μιας τέτοιας κατάστασης σε μία χώρα να μπορεί να προστατευτεί και στην άλλη. Δεν αφορούν μόνο τα θύματα ε, βίας λόγω διακρίσεων, λόγω του φύλου για παράδειγμα. Υπάρχουν και τα παιδιά Υπάρχουν ε, πολλοί άνθρωποι, όπως για παράδειγμα οι, οι whistleblowers για παράδειγμα, που πολλές φορές επίσης διώκονται. Ευχαριστώ η κυρία Παρβανόβα. Πολύ σύντομα, πολύ σύντομα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Άρχισα να αναρωτιέμαι, όταν μιλάμε για άντρες που είναι άντρες, είναι ποινικό όταν ε, ένας άντρας ε, ε, δέρνει μια γυναίκα είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για μένα... Για μένα η διάκριση που γίνεται στη μεταχείριση ήδη είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τα ίδια πρότυπα και εάν προστατεύουμε τα κεφάλαιά μας ή τις επιχειρήσεις μας όταν μεταφέρονται από ένα κράτος μέλος σε κάποιο άλλο, τότε θα πρέπει να ισχύει για το ίδιο μας το σώμα. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ, έχουμε πολύ λίγο χρόνο. Ένα λεπτό για το Συμβούλιο, την Κομισιόν και μια εισηγήτρια. Πρώτα, τον λόγο στον ε, ε, εκπρόσωπο του Συμβουλίου. Παρακαλώ. Ε, Θα είμαι πολύ γρήγορος. Η Κομισιόν λέει ότι έχουμε δύο μηχανισμούς, έναν ποινικό, έναν αστικό. Αυτό είναι αδύνατον, γιατί λέμε στο θύμα, τι λέμε, ότι θα έχετε χώρες με ποινικό σύστημα και χώρες με αστικό, μα το θύμα μπορεί να μετακινηθεί από όπου θέλει σε όπου θέλει. Δεν μπορεί αλλού να υπάρχουν αστικά μέτρα και αλλού ποινικά. Θα πρέπει να συνδυαστούν αυτά τα δύο συστήματα. Είναι απολύτως αναγκαίο. Πώς μπορούμε να πούμε σε ένα ε, θύμα «Α, αν πάτε από τη Γερμανία στην Αυστρία έχει καλώς, αν πάτε από τη Γερμανία στην Ισπανία δεν ισχύει το σύστημα». Είναι αδιανόητο. Θα πρέπει να συνδυάσουμε τα δύο μέσα. Και το μόνο αδίκημα της Ισπανικής ε, Προεδρίας ήταν που υπέβαλε αυτή την πρόταση. Η προηγούμενη Κομισιόν συμφωνούσε και στην ουσία ήταν μια διελκυστίνδα εξουσιών μεταξύ Κομισιών και συμβουλή. Η, η Ισπανική Προεδρία κατέβαλε κάθε προσπάθεια προσέγγισης με την Κομισιόν με την τελευταία πρόταση. Αλλά η Κομισιόν δεν δέχτηκε αυτό το νομικό πλαίσιο. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούσαμε. Μιλάμε για όλα τα θύματα. Όλα, όλα. αλλά στην πλειοψηφία πρόκειται για οικιακή βία. Μιλάμε όμως για όλα τα θύματα. 12 κράτη-μέλη υπέβαλαν αυτή την πρόταση. Ευτυχώς μας υποστηρίζουν περισσότερα κράτη από 12. Η αρχική πρόταση όμως ε, έγινε από 12 κράτη. Και τέλος, θα ήθελα να πω ότι αυτά θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε έναν μελλοντικό μηχανισμό. Ελπίζω η Κομισιόν να τον παρουσιάσει το 2011, γιατί πρόκειται για ένα ευρύτερο ζήτημα το οποίο θα οδηγήσει σε μεγάλες συζητήσεις. Ας κάνουμε το πρώτο βήμα και εάν είναι ελληματικό θα το επιλύσουμε μαζί. Αφήστε μας όμως να το επιλύσουμε. Δεν θα μπω στο 9 σε. Αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε. Αλλά Ας κάνουμε αυτό, ας το συζητήσουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Κομισιόν. Κύριε Φάουλ, παρακαλώ. Right, um, Ένα λεπτό. Θα είμαι πολύ σύντομος. Στις 25 Μαΐου θα γίνει συνάντηση με εμπειρογνώμονες από τα κράτη-μέλη για να συζητήσουμε όλα τα θέματα αυτά και θα είμαστε ε, ευχαριστημένοι αν η Κομισιόν, εάν το Κοινοβούλιο στείλει εκπροσώπους στη συνάντηση αυτή. Εδώ το θέμα δεν είναι η διελκυστίνδα. Όποιο όμω και να πάρει την πρωτοβουλία, η Κομισιόν ή το Συμβούλιο, θα πρέπει να είναι σωστό ο νόμο που θα προκύψει. Αλλιώ θα καταρρεύσει και δεν το θέλουμε αυτό, διότι αυτό θα ε, ζημιώσει την ε, εικόνα όλης της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Φυσικά είναι ε, παραβίαση των θεμελιωτών δικαιωμάτων το να ε, ασκεί κανεί σε βία σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Αλλά η συνθήκη δεν προβλέπει νομική βάση για την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Μόνο η συνθήκη το κάνει αυτό. Και η συνθήκη είτε μας αρέσει είτε όχι κάνει τη διάκριση ανάμεσα στο, αστικό δίκαιο και στο ποινικό δίκαιο. Δεν την συνέγραψα εγώ τη συνθήκη μπορώ μόνο να την εφαρμόζω ως έχει. Είναι δουλειά της Κομισιόν ως θεματοφύλακα των συνθηκών να σας προειδοποιεί ότι αυτή είναι η κατάσταση. Έχετε μια νομική υπηρεσία, ακούστε την γνωμοδότησή της. Ε, εάν εμπιστεύομαι εγώ τη γνωμοδότηση της νομική μου υπηρεσίας. Ε, ε, περιμένω να γίνει σεβαστή και από άλλους. Θέλουμε λοιπόν μια σωστή πρόταση με σωστή νομική βάση, σωστή προετοιμασία, σωστή διαβούλευση, σωστή ανάλυση. Θα πρέπει να γίνουν διαβουλεύσεις με όλους. Θα πρέπει να υιοθετηθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και να καλύπτει όλες τις πιθανές χρήσεις μιας ευρωπαϊκής προστασίας εντολής. Θα έχει μόνο μερική ε, μερικό αποτέλεσμα και έτσι δεν θα είναι ικανοποιητική. Ε, δεν είναι δύσκολο το θέμα. Ε, δεν έχει να κάνει με κανένα πόλεμο και λυπάμαι πάρα πολύ που αναφέρθηκε το θέμα αυτό. Δεν πιστεύω ότι είναι η κατάλληλη λέξη σε περίπτωση. Η συνθήκη παρέχει τρία διαφορετικά άρθρα, 82 για το ποινικό δίκαιο, 84 για την πρόληψη εγκλημάτων που έχει αναφερθεί αλλά δεν καλύπτεται, λυπάμαι, από την πρόταση. Δεν μπορεί να καλύπτεται διότι δεν υπάρχει απαραίτητη νομική βάση και το αστικό δίκαιο είναι ξεχωριστό. Άλλα κράτη-μέλη εμπλέκονται, η Δανία θα συμμετέχει σε ένα αλλά όχι σε άλλα. Η... Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία θα έχουν opt-in, θα έχουν δυνατότητα συμμετοχή για το ένα μέσο και όχι για το άλλο. Ε, και τελικά τι θα έχουμε, patchwork θα έχουμε και κατακαιρματισμό. Δεν θέλουμε αυτό να προσφέρουμε στα θύματα της βίας αξίζουν κάτι καλύτερο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Χιμένες. Ένα λεπτό. Και στην κυρία Ρομέρο. Ένα λεπτό. Παρακαλώ, κυρία Χιμένες. Ε, Θα είμαι πολύ σύντομη. Αρχίσαμε ακούγοντας και επειδή το οφείλουμε στα θύματα θα πρέπει οι εισηγήτριες, το Συμβούλιο και η Κομισιόν να σκεφτούμε. Να σκεφτούμε τι ακούσαμε, πρέπει να μελετήσουμε, να περιμένουμε μέχρι την 4η Ιουνίου που θα μας υποβληθεί το κείμενο, να δούμε κατά πόσο θα συμφωνήσει το Συμβούλιο και να έχουμε μια καλή βάση ανεξάρτητα ανεξάρτητα από το κατά πόσο θα προβάλλουμε τροπολογίες ή όχι. Θα πρέπει να έχουμε μία σωστή βάση. Δεν θέλω να δώσω στα θύματα φρούδες ελπίδες. Δεν θέλω να γίνει αυτή η δόλια μεταχείριση του θύματος, των θυμάτων. Ας σκεφτούμε τι ακούσαμε γιατί όλοι έχουν εν μέρη δίκιο και με το χρόνο που έχουμε μπροστά μας θα φτάσουμε στην καλύτερη δυνατή λύση. Το ελπίζω εκ βάθους καρδίας. Ευχαριστώ κυρία Ρομέρο, παρακαλώ. Ελπίζω το Κοινοβούλιο να διαμεσολαβήσει έτσι ώστε να αρθούν τα ερωτηματικά. Δεν είναι η πρώτη φορά που η νομική υπηρεσία της Επιτροπής διαφέρει από την άποψη της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου. Δηλαδή έρχονται σε σύγκρουση διάφορες νομικές υπηρεσίες. Υπάρχει απόκληση. Τώρα όμως θα πρέπει να εργαστεί το Κοινοβούλιο, να μπει επί της ουσίας και με την διαμεσολάβηση του Κοινοβουλίου θα δούμε πώς θα επιλύσουμε ένα θέμα που σίγουρα μπορεί να επιληθεί. Διότι όταν, όπου υπάρχει θέληση ε, είμαι ε, πεπισμένη ότι θα επιληθεί το ζήτημα και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για ε, θύματα μιας τέτοιας ανεπίτρεπτης βίας. Ευχαριστώ θερμά όλους τους συμμετέχοντες στην Κομισιόν, το Συμβούλιο, την Επιτροπή Λύπε που συμμετείχε τόσο ενεργητικά στο θέμα αυτό. Θα επανέλθουμε στη συνέχεια της συζήτησης, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, στις 31 ε, Μαΐου, όπου η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θα οργανώσει κοινή συζήτηση μαζί μας. Είμαι πεπισμένη ότι θα προοδεύσουμε στο θέμα αυτό, προς όφελος όλων των θυμάτων αυτής της βίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αύριο 9 η ώρα το πρωί. Μην ξεχάσετε, βρισκόμαστε σε άλλη αίθουσα. Πάρτε μαζί σας όλα τα έγγραφά σας. Σας ευχαριστώ πολύ.